So, dear colleagues, uh, I propose that we start. Uh, I Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω να σας κάνω κάποιες ε, ανακοινώσεις. Ε, σήμερα το πρωί η κυρία Ρέκνερ ορίστηκε ε, εισηγήτρια για την άρση ασυλίας του κυρίου Ζαμαρή Λεπέν και ο κύριος Χρυσόχρονος εισηγητής για την άρση ασυλίας του κυρίου Ζαν Φρανσουά κύριος Βιέφκα για τους ε, αφαιρέγγιους. Ε, επίσης έχουμε ένα ψήφισμα που κατατέθη από τον κύριο, σε σύμφωνία με τον κανονισμό 133 του καταστατικού όσον αφορά τις πόλεις της περιφέρειας του Βένετο για εμπορικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις μη ευρωπαϊκές χώρες και από τον Ντομινίκ Μαρτέν για την επιτάχυνση των πληρωμών. κ. Ναγκρέσκου θα συμμετάσχει στο φόρουμ για την εσωτερική διακυβέρνηση. Τέλο, ο κ. Κανιέτα θα κληθεί να παρακολουθεί στη συνεδρίαση τη Επιτροπή ε, ε, Νομικών Υποθέσεων στι 12 Ιουλίου 2016. Yes, I, I, uh, I uh, welcome Καλώς ορίζω την Επιτροπή και θα δώσω το λόγο στους εκπρόσωπους της Γενικής Διεύθυνσης για την Οικονομική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιογορών. Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε εσάς και τα πορίσματα στα οποία καταλήξατε μετά από τη δημόσια διαβούλευση για τις μη δεσμευτικές κατευθυντήρες γραμμές. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να έρθουμε στην Επιτροπή σας για να σας ενημερώσουμε σε σχέση με τα πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης για τις μελλοντικέ μη δεσμευτικές γραμμές για τη διευκόλυνση των μη της, της, εφαρμογής ε, των αναφορών για τις ε, μη χρηματοπιστωτικές ε, υποχρεώσεις. Ε, η διαβούλευση ε, τελείωσε πριν από λίγους μήνες και έχουμε πολλά σχόλια. Δεν δημοσιεύσαμε ακόμα τη δήλωση feedback πορισμάτων, το προετοιμάζουμε, αλλά με χαρά θα μοιραστούμε μαζί σας ήδη ως πρώτο πιάτο ε, τα προκαταρκτικά μας πορίσματα. Θα αρχίσουμε τη σύνταξη και των κατευθυντηρίων γραμμών βεβαίως. όπως προβλέπετε, για την δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Θα δώσω το λόγο στον Νικολά Μπερνιέ που θα σας ενημερώσει για τα προκαταρκτικά αυτά απορίσματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα θέλαμε σήμερα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσουμε την ε, σύνοψη των ευρημάτων μας. Okay, yes. Um, first of all, uh, remind you that... Καταρχάς, ε, να σας θυμίσω ότι η δουλειά που κάνουμε τώρα όσον αφορά την εκπόνηση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών ε, βασίζεται στην οδηγία 2014-95 ε, ε, για την κοινοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλους ομίλους. Τα κράτη-μέλη ακόμα εφαρμόζουν την διαδικασία αυτή στην ε, εθνική νομοθεσία. Αυτό θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2016 και η Κομισιόν έχει οργανώσει ανεπίσημα σεμινάρια με εκπροσώπου των κρατών μελών για να διευκολύνει την ε, διαδικασία της μεταφορά. Ε, Τρει συναντήσει είχαμε μέχρι τώρα, την πρώτη τον Φεβρουάριο του 2015 και τον Σεπτέμβριο του 2015 και έχουμε προγραμματίσει άλλη μία φέτος. Το πιθανότερο είναι φέτος τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να πραγματοποιηθεί τελευταία. Το άρθρο 2 της οδηγίας ε, προβλέπει ότι η Κομισιόν θα, θα προετοιμάσει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία για την κοινοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Φέτος τον Ιανουάριο ξεκινήσαμε δημόσια διαβούλευση που διήρκησε μέχρι τα μέσα Απριλίου. Ουσιαστικά ζητήσαμε ε, την άποψη ενδιαφερομένων μερών ε, σχετικά με το σε ποιον απευθύνονται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τι στοιχεία κάνουν πιο χρήσιμες ε, και πιο επίκαιρε τις πληροφορίες αυτές και κατά τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών είναι προτιμητέα μια γενικότερη λύση όσον αφορά τις γενικές αρχές. Επίσης ρωτήσαμε σχετικά με τους κύριους δείκτες επιδόσεων. καθώς και την σχέση ανάμεσα στις κατευθυντήρες γραμμές και άλλα εθνικά και διεθνή πλαίσια. Και επίσης ρωτήσαμε κατά πόσο θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνονται διάφορες ε, άλλες ε, πληροφορίες, πληροφορίες για την πολυμορφία. Λάβαμε συνολικά 355 απαντήσεις. πολύ περισσότερες, δηλαδή από όσες λάβαμε το 2010 κατά την διαβούλευση για την ίδια την οδηγία. Τότε είχαμε λάβει 259 απαντήσεις. Αυτό πιστεύουμε ότι δείχνει αναγνώριση των ενδιαφερομένων μερών, ε, επενδυτών, επιχειρήσεων κλπ Ε, σχετικά με τη σημασία των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των πληροφοριών για την πολυμορφία και για τις μη δεσμευτικές κατευθυντήρες γραμμές. Επίσης, ε, είναι ε, αρκετά διαφορετικές οι απαντήσεις που έχουμε λάβει και πιστεύουμε ότι καλύπτουν όλο το σκηνικό και όσον αφορά την συμμετοχή των διαφορών ειδών ενδιαφερομένων μερών, ε, καθώς και όσον αφορά την γεωγραφική ισορροπία. Βλέπετε εδώ στην εικόνα ότι πολλές απαντήσεις ε, έχουν ε, παραλυφθεί από επιχειρήσεις και οργανώσεις επιχειρηματιών. Πολλές προέρχονται από μη κυβερνητικέ οργανώσει και την κοινωνία των πολιτών, περίπου το 1 τέταρτο. Και επίση έχουμε λάβει απαντήσει από ελεγκτές, λογιστές και άλλου επαγγελματίες, από δημόσιες αρχές, καθώς και από άτομα, από ιδιώτες. Όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία, βλέπετε ότι έχουμε λάβει απαντήσεις από πολλά κράτη-μέλη. Πάνω από 50 ήταν Ε, γερμανικές. Επίσης από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο λάβαμε πολλές, πάνω από 30. Λάβαμε και απαντήσεις από ευρωπαϊκούς οργανισμούς που εδρεύουν στις Βρυξέλλες. Επίσης, λάβαμε σημαντικό αριθμό απαντήσεων από μικρά κράτη-μέλη και από τρίτες χώρες επίσης. Όπως ανέφερα ήδη, σχεδόν το μισό των απαντήσεων προέρχονταν από επιχειρήσεις και ε, οργανώσεις ε, επιχειρηματιών, εργοδοτών. Και πιστεύουμε ότι οι απαντήσεις που έχουμε λάβει παρουσιάζουν με τρόπο τις απόψεις των επιχειρήσεων που θα καλύπτονται από την νομοθεσία αυτή καθώς και από τις κατευθυντικές γραμμές που θα ακολουθήσουν. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση δηλώνουν ότι κοινοποιούν κάθε χρόνο μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Οι επιχειρήσεις αυτές λοιπόν έχουν ήδη την τεχνογνωσία και εμπειρίες. Γνωρίζουν τι χρειάζεται για να παρέχονται αυτές οι πληροφορίες και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κοινοποίησης. Οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούν ήδη υπάρχοντα πλαίσια υποβολής εκθέσεων. Δυστυχώς ε, είναι περιορισμένα αυτά που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα. Αυτό όμως ε, που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από πλευρά των ενδιαφερομένων, από όλες τις κατηγορίες τους, Ε, για την σημαντικότητα των πληροφοριών, το materiality. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ε, ότι είναι σημαντικό στοιχείο αυτό και ότι οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες στις μη κατευθυντικές γραμμές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη σημαντικότητα και την επικαιρότητα, τη χρησιμότητα των πληροφοριών αυτών. Θα πρέπει δηλαδή να κοινοποιούνται πληροφορίες χρήσιμες ε, και όχι άλλες. Και μάλιστα να μην ε, είναι υποχρεωτική δημοσίευση άλλων πληροφοριών. Άλλα στοιχεία είναι η χρησιμότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών. Και άλλες και που δεν τονίστηκαν εξίσου από τους ε, ενδιαφερομένους είναι η συγκρισιμότητα και η αποφυγή ε, περί του γραφειοκρατικού άχθους. Άλλο σημαντικό στοιχείο για μας είναι το πώς οι κατευθυντήριες γραμμές ε, θα πρέπει να ε, χειρίζονται τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Οι περισσότερες απαντήσεις έλεγαν ότι προτιμητέο είναι να παρουσιάζονται οι γενικές αρχές, ενώ περίπου το 1 τρίτο ήθελαν πιο αναλυτική προσέγγιση όσον αφορά την εκπόνηση των κατευθυντήριων γραμμών. Επίσης, ρωτήσαμε σχετικά ε, με ε, τους κύριους δείκτες επιδόσεων και τις ποσοτικοποιημένες πληροφορίες. Αναλύοντας τις απαντήσεις διαπιστώσαμε ότι υπάρχει προτίμηση για ευελιξία, για Νομίζω ότι έτσι σας έδωσα μία γενική επισκόπηση σύντομη ε, των πληροφοριών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εντός κάποιων εβδομάδων οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα μας και υπολογίζουμε να ολοκληρωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές μας μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα χαρώ να ακούσω τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Δίνω τον λόγο στους ευρωβουλευτές, εάν έχουν ερωτήσεις. Σέζιο, παρακαλώ. Κοφαγάτη. Ευχαριστώ. Κάνατε πολύ σημαντική εργασία. Νομίζω πως αντικειμενικά αποτελεί μια συμβολή, κατά τη γνώμη μου, αξιόλογη. Να εισάγονται οι μορφές διαφάνειας που αφορούν την οικονομία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, παλαιότερα εργαστήκαμε πολύ και πολύ αποφασιστικά εδώ σε αυτή την Επιτροπή και όχι μόνο, ώστε να φτάσουμε σε ε, συμπεράσματα όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για την ε, δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών που έχουν σημαντικές, ε, για στοιχεία που έχουν σημαντικές επιπτώσεις για συγκεκριμένους τομείς. Εκτιμώ το πνεύμα για τις προθέσεις σας. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές που δεν είναι δεσμευτικές ε, κατά την άποψη της Επιτροπής πώς ε, θα υποστηριχτούν ε, από την συγκρισιμότητα με τις πληροφορίες που καλούνται να δίνουν οι, μικρ... οι μεμονωμένες επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζουμε τις προθέσεις της κάθε εταιρείας, αλλά να τις συγκρίνουμε με ε, τις πληροφορίες άλλων αντίστοιχων εταιρεών. Πώς λοιπόν η Κομισιόνα θα μπορέσει να εγγύθει ότι θα μπορούμε να συγκρίνουμε α, να, τις, τις ε, διάφορες αυτές κατευθύνες γραμμές. Έπειτα, αναφερόμενα στην οδηγία που εγκρίθηκε Αυτές οι κατευθυντήριε γραμμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ε, δείκτες ε, παροχών, τομεκές και ένα εταιρεία. Έτσι λέει το κείμενο. Το Ευρωκοινοβούλιο στη συζήτηση που κάναμε πριν την ψηφοφορία επανειλημμένα είχαμε πει ότι αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά όχι μόνο για τη δυνατότητα σύγκρισης που έλεγα προηγουμένως, σύγκριση ανάμεσα στις ε, πληροφορίες που δίνουν οι διάφορες επιχειρήσεις, αλλά ήταν σημαντικές ε, γιατί ε, μπορούμε έτσι να εντοπίσουμε συγκεκριμένα ποιες θα είναι ακριβώς αυτοί οι δείκτες, αυτές οι πληροφορίες. Γιατί είναι προφανές ότι στη συνολική αξιολόγηση υπάρχουν δείκτες οι οποίοι έχουν διαφορετική αξία μεταξύ τους. Υπάρχουν αυτοί που είναι οικονομικού χαρακτήρα ε, και αυτοί που είναι κοινωνικού χαρακτήρα και που καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτούς τους πρώτους δείκτες. Θα σας ήμουν λοιπόν ευγνώμων αν θέλατε να μας δώσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με αυτό το πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει η εργασία μας. Σας ευχαριστώ. Merci, Monsieur Durand. Ευχαριστούμε. Ο κ. Durand. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά το Σέργιο Κοφεράτη δυσκολεύομαι να λάβω το λόγο γιατί είναι πολύ εξυπνότερο σε μου και καταφέρνει να κατανοήσει μέσω των δηλώσεών σας κάτι που εγώ δεν κατανόησα. Δηλαδή, το συγγνώμη, εγώ φταίω, σίγουρα, αλλά δεν κατάλαβα ποια κριτήρια οδήγησαν σε αυτό τον οδηγό. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα, τι είδου ζητήματα, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, δεν ξέρω τι άλλο, τι θέματα συζητήσατε με τις επιχειρήσεις και με όλους αυτούς που απάντησαν στις ερωτήσεις. Άκουσα, συγγνώμη που το λέω, γενικότητες, αλλά δεν κατάλαβα το συγκεκριμένο θέμα επί του οποίου ετέθησαν οι ερωτήσεις. Αυτά ζητώ συγγνώμη που δείχνω απλοϊκός, αλλά προς το παρόν δεν έχω καταλάβει. Πρόεδρος. Κύριε Τιουχόμ, ίσως δεν είστε ο μόνος, αλλά είμαι βεβαία ότι η Επιτροπή θα μας δώσει λεπτομέρειες, πιο συγκεκριμένα στοιχεία για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Δίνω το λόγο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Όπως είπαμε, πρόκειται για μια ε, δημόσια διαβούλευση που έγινε επί τρεις μήνες και όλα τα ερωτήματα ε, δημοσιεύθηκαν. Και αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία τα οποία αποκομίσαμε από την διαβούλευση. Δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει πώς θα συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί καν το feedback που έχουμε πάρει από το ερωτηματολόγιο, από τη διαβούλευση. Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία και απλώς σας αναφέρουμε τα πρώτα μας ευρήματα. Δεν έχω κι εγώ να σας πω τίποτα παραπάνω στο στάδιο αυτό. Δεν έχουμε καν ολοκληρώσει τη συζήτηση σε εσωτερικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ε, παρουσίαση που κάναμε σε PowerPoint ε, είδατε κάποια στοιχεία. Κάποιες ε, απαντήσεις δείχνουν ότι πρέπει να παραμείνουμε στις γενικές αρχές και οι δείκτες απόδοσης δεν θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ άλλες απαντήσεις προτείνουν να προχωρήσουμε περισσότερο σε κάποιους τομείς. Δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει την Επιτροπή και δεν μπορώ να σας πω τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Δώστε μας λίγες εβδομάδες τουλάχιστον για να το επεξεργαστούμε και με τα χαράς να επανέλθω στην Επιτροπή σας και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες αφού πρώτα κάνουμε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Και για την ερώτηση του κυρίου Κοφεράτη, λέει η Πρόεδρος, δεν έχετε απάντηση προς το παρόν. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Ευχαρίστω να απαντήσω, αλλά είμαστε σε τόσο προκατακτικό στάδιο της ανάλυσης που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ωραία, δεν θα επιμείνουμε, λέει η Πρόεδρος. Ελπίζουμε ότι σε μια μεταγενέστερη συνεδρίαση θα έχετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία να μας δώσετε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κοφεράτη ζητά το λόγο. Σημειώνω ότι δεν αρκεί η καλή θέληση αλλά μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε μία ένδειξη χρονική για το πότε θα μπορέσετε να μας δώσετε κάποιες καταληκτικές απαντήσεις γιατί ακόμα μια τέτοια ακρόαση θα την απέφευγα. Μάλιστα κύριε Κομφεράτη. Ευχαρίστω θα επανέλθουμε αμέσω μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ, δηλαδή αρχέ Σεπτεμβρίου. Okay, we will take note uh, no, but it's good that. Uh, Μάλιστα, το σημειώνουμε. Όχι, καλό είναι. Κάποια δουλεύουν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Λίγα λεπτά διάλειμμα για να καταφτάσουν οι προσκεκλημένοι για την ακρόαση για την Ουκρανία. Dear colleagues, let us begin. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε. Καλωσορίζω τους προσκεκλισμένους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την ακρόαση για την ε, μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ουκρανία οργανώνεται από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και την αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική συνέλευση Euronest. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Πετρέγκο, αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου κυρία Σιρόιντ, Γενικό Εισαγγελέα Λουτσέγκο και την Επίτροπο Βέρα Γιούροβα, μεταξύ πολλών άλλων διακεκριμένων προσκεκλημένων ιδιαίτερα από την Ουκρανία. Ο κύριος Πετρέγκο συνοδεύεται από τον κύριο Γιάντσου, αναπληρωτή Υπουργό δικαιοσύνη. Και ο Γενικός Εισαγγελέας συνοδεύεται από τον κύριο Ιδιαίνη Γέννη, αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα. Μετά τις εισαγωγικές παρατηρήσεις θα οργανωθούν δύο συζητήσεις. Η πρώτη συζήτηση θα ασχοληθεί με την μεταρρύθμιση του συντάγματος και του δικαστικού σώματος και οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν από μια παρέμβαση της κυρίας Χάουταλα, συμπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest και μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. και θέματα σχετικά με το στάτους των δικαστικών. Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο πέρυσι επισκέφθηκε το Κίεβο. Η σημερινή ακρόαση αποτελεί συνέχεια των συναντήσεων που κάναμε στο Κίεβο θέματα που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Είχαμε κάνει συναντήσεις ε, με το Κοινοβούλιο, την Βαρχαούνα Ράντα, τον πρόεδρο Ποροσέγκο, ε, μονάδες για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, μονάδα κατά της διαφθοράς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα, ένα πιο πρακτικό ζήτημα. Ξέρετε ότι ο χρόνος είναι χρήμα στο Κοινοβούλιο και ζητώ συγνώμη που θα πρέπει να σας αστυνομεύω λίγο όσον αφορά το χρόνο. Δίνω το λόγο στον Αντρέη Πλέγκοβιτς, επικεφαλής Τη αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανία. Πολύ σύντομη όμως ε, παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ Παύλ, κυρία Επίτροπε, κύριε Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που οργανώνεται εδώ από κοινού από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και την Αντιπροσωπή για τις σχέσεις με την Ουκρανία της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος και πιστεύω ότι είναι μια ε, ιδιαίτερα επίκαιρη προσέγγιση από την Νομική Επιτροπή, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου ε, για να τονίσουμε τη σημασία που έχουν οι μεταρρυθμίσεις του δικαστικού τομέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευρύτερη ευρωπαϊκή ε, ατζέντα της Ουκρανίας Ιδίω ε, και εν ώψη των συζητήσεων για απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίου. Ε, προσβλέπω σε μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Θέλουμε να ακούσουμε τι έχουν να μα πούν και οι Ουκρανοί συνάδελφοι από τη δική του εμπειρία και γύρω στι 6 το απόγευμα θα προσπαθήσω να κλείσω με τη δική μου παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Βέρα Γιούροβα. Ευχαριστώ κύριε Σβόμποτα, ε, αγαπητοί συνάδελφοι ε, και προσκεκλημένοι από την Ουκρανία. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ για, την, ε, για το πόσο επίκαιρη είναι αυτή η ακρόαση. Σήμερα έχουμε εδώ σημαντικούς παράγοντες για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της Ουκρανίας. Κάτι που μας δημιουργεί ελπίδες για μια πολύ χρήσιμη και επικοδομητική συζήτηση. Περιμένω να ακούσω από εσάς εδώ και από τους συναδέλφους από την Ουκρανία τις εξελίξεις και τις προβλέψεις για το εγγύς μέλλον. Σήμερα βρίσκομαι εδώ ως φίλη της Ουκρανίας και θα ήθελα να συμβάλλουμε στην συνεχιζόμενη εφαρμογή ε, επιτυχών μεταρρυθμίσεων. Επισκέφθηκα την Ουκρανία για να δω εγώ ίδια την κατάσταση και να τη συζητήσω με τις αρχές, ε, με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με τη διεθνή κοινότητα που παρέχει συμβουλές ε, και υποστήριξη. Επί πολλά χρόνια η έχει αναγνωριστεί η μεταρρύθμιση του δικαστικού ως ε, μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προτεραιότητες στην ε, Ουκρανία. Ε, ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και θα επιτρέψει στους πολίτες της Ουκρανίας να εμπιστεύονται το κράτος τους. Σε ιστορικό χαμηλό είχε φτάσει ε, η εμπιστοσύνη του κοινού στο δικαστικό σύστημα και υπάρχει ε, γενική απέτηση για μεταρρύθμιση. Γι' αυτό Χαίρομαι που το παρόν κοινοβούλιο και η παρούσα κυβέρνηση έχουν ε, λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Τον Ιούνιο υιοθετή... Στις 2 Ιουνίου υιοθετήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις, όπως μόλις μας είπε ο κύριος Σβόποτα. Είναι σημαντικό βήμα αυτό για να ευθυγραμμιστεί απόλυτα το δικαστικό σύστημα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του από κυβερνητικές επιρροές. Τώρα θα πρέπει να ε, δώσουμε έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων ε, για να πετύχουμε αποτελέσματα στην πράξη, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των Ουκρανών ε, για ένα ανεξάρτητο, αποτελεσματικό και υψηλής ποιότητας δικαστικό σύστημα. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις δείχνουν κοινή κατανόηση ότι πρέπει να υπάρχει ακαιρεότητα. Για να υπάρχει εμπιστοσύνη προς το δικαστικό σύστημα, κάθε δικαστής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος και να ε, μην υφίσταται εξωτερικές πιέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θεωρούνται όλοι οι δικαστές αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι, ώστε το κοινό να ε, έχει εμπιστοσύνη ότι θα ε, κριθεί δίκαια η υπόθεσή του. Θα πρέπει λοιπόν να επικροτήσουμε την προσπάθεια για την Επιτροπή Αξιολόγησης των Δικαστών, ε, παρότι ε, θα πρέπει να βελτιωθεί η δουλειά με καλύτερους ε, ελέγχους. Επίσης θα πρέπει να είναι διαφανείς οι διαδικασίες διορισμού και προαγωγής. Και επίσης θα πρέπει να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών. Για όλα λοιπόν τα θέματα αυτά είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα θίξει εδώ το πρώτο πάνελ μας. Χαιρόμαστε που έχουμε εδώ στο πάνελ μας εκπροσώπους και των τριών βασικών τομέων του κράτους καθώς και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η μεταρρύθμιση της εισαγγελία επίσης αποτελεί προτεραιότητα για την, Τουρκία, για την Ουκρανία και χαίρομαι που ο νεοδιοριστής ε, Γενικός Αγγελέας κ. Ζουτσέγκο ε, θα συζητήσει εδώ μαζί μας σήμερα το μέλλον ε, του, του συστήματος εισαγγελέων. Σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την μεταρρύθμιση του συστήματος επιβολής του νόμου και του δικαστικού συστήματος της Ουκρανίας και περιμένω ενδιαφέρον να ακούσω τα αποτελέσματα της σημερινής σας συζήτησης. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία ε, στην συνέχιση των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ο πρέσβης κύριος Τομπίνσκι. Πέντε λεπτά μόνο. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, Πρόεδρε των Διαφόρων Επιτροπών. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κίεβο από το Σεπτέμβριο του 2012. Δεν θυμάμαι κανένα δημόσιο πρόσωπο στην Ουκρανία που να ισχυρίζεται ότι λειτουργούν σωστά το σύστημα δικαιοσύνης ε, και το κράτος δικαίου στην Ουκρανία. Είναι ένα γνώρισμα του ουκρανικού συστήματος το οποίο επί δεκαετίες ίσχυε. Και το αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης στο δικαστικό σύστημα στην Ουκρανία, όπως ανέφερε και η Επίτροπος, γιατί μόνο 5% εμπιστοσύνη υπάρχει, ε, είχε επίπτωση και στην εμπιστοσύνη στο κράτος συνολικότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλους εταίρους προσπάθησε να βελτιώσει την Ουκρανία, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις ελλείψεις του συστήματος. Ο κύριος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, που μας βοηθά να υλοποιήσουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις, να αξιολογήσουμε κάποιες διατάξεις, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει από μόνη της κοινοτικό κεκτημένο για το πώς να δημιουργήσει ένα σύστημα δικαστικό και θεσμικό για την ε, ε, επιβολή του δικαίου και για τα δικαστήρια γενικότερα στην Ουκρανία. Το Συμβουλίο της Ευρώπης ε, μας βοηθά σε αυτό το τομέα γιατί ε, μπορούμε έτσι να συγκρίνουμε το σύστημα στην Ουκρανία με διεθνείς ε, συνθήκες και συμβάσεις. Να σας πω τι κάναμε τα τελευταία χρόνια. Υλοποιήσαμε κάποια προγράμματα βοήθειας και το κύριο πρόγραμμα με το οποίο είχαμε ξεκινήσει πριν από την επανάσταση του φθινοπόρου του 2013 είναι το πρόγραμμα υποστήριξης ε, για μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα στην Ουκρανία. Το πρόγραμμα αυτό δεν το έβλεπαν με πολύ καλό μάτι οι προηγούμενες αρχές και η πολιτική ελίτ της Ουκρανίας και το υιοθέτησε ο νέος Υπουργός που ε, ανέλαβε καθήκοντα μετά την ε, επανάσταση της αξιοπρέπειας και προσπάθησε να περάσουν τις μεταρρυθμίσεις για όλους τους θεσμούς, ούτως ώστε να υπάρχει μια οριζόντια καθοδήγηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι ε, τμήμα μιας συστηματικής μεταρρύθμισης της Ουκρανίας με οριζόντια, με οριζόντιες κατευθύνσεις και ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε οριζόντια υποβοήθηση και κατευθύνσεις. Προσπαθήσαμε λοιπόν ε, να δώσουμε κατευθύνσεις για διαφορετικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις δομές. και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε να εξηγενθεί η πολιτική στο δικαστικό τομέα, μια πολιτική που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο της Ευρώπης και μετά την Επανάσταση του 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδίασε ένα συμβόλαιο ε, με πολλαπλά στοιχεία που συμπεριλάμβανε και την ε, μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος ώστε να γίνει διαφανές και αμερόληπτο και να το βλέπουν έτσι και οι πολίτες της Ουκρανίας. Η υλοποίηση αυτού του συμβολέου έχει άμεση σχέση με το πρόσφατα υιοθετηθέν ε, Σύνταγμα της Ουκρανίας και με το σύστημα υλοποίησης για τα δικαστήρια και για το δικαστικό σώμα στην Ουκρανία. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε και μια συμβουλευτική αποστολή στην Ουκρανία και ο επικεφαλής της συμβουλευτικής αυτής αποστολής θα λάβει το λόγο για να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη δουλειά που γίνεται επί τόπου για να βοηθήσουμε τα θεσμικά όργανα στην Ουκρανία ώστε να υλοποιήσουν στην πράξη τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά την αστυνομία, αλλά και για να ελέγχουν έχουν ε, την τήρηση των ε, δικονομικών κανόνων ε, στην Ουκρανία. Ένα μεγάλο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης, δίνοντας έμφαση σε ένα σημείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί συστημικά στην Ουκρανία. Όλα αυτά συνδέονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί η διαφθορά δεν είναι μόνο ηλική, είναι διαφθορά της κουλτούρας γενικότερα και διαφθείρει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος. Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε δεν είναι μόνο η φιλία μας προς την Ουκρανία, αλλά και γιατί είναι προς συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν μια γειτονική μας χώρα, σχεδόν η μεγαλύτερη γειτονική μας χώρα, είναι μια χώρα που έχει ένα σύστημα δικαιοσύνης που λειτουργεί σωστά, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν, που επιτρέπει στο εμπόριο να λειτουργεί, που επιτρέπει την προστασία όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν από και προς την Ουκρανία και που μας ε, διασφαλίζει ότι λειτουργεί σωστά ο κρατικός μηχανισμός. Όλα αυτά αποτελούν το κλειδί για τη μεταρρύθμιση όλων των άλλων τομέων στην Ουκρανία και για να δημιουργηθεί η βάση για την οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε λεπτά ακριβώς μίλησα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Έλμαρ Μπρόκ πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Για πέντε λεπτά με τη στενή έννοια. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα το ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, έχει οργανώσει την ε, σημερινή συνάντηση για να διαπιστωθούν οι πρόοδοι. Θυμάστε πριν δύο χρόνια το κίνημα Ευρωμαϊντάν και ένα από τα βασικά αιτήματα τότε ήταν ε, ένα δίκαιο δικαστικό σύστημα. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της επανάστασης της αξιοπρέπειας. Το να υπάρχει δίκαιο δικαστικό σύστημα. Από την άλλη μεριά, βλέπω πόσο δύσκολο είναι να μεταρρυθμίσει κανείς σε μια εμπόλεμη χώρα. Τη στιγμή που παραβιάζεται η εδαφική ακαιρεότητα μιας χώρας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν ε, πολιτικές, ε, οικονομικές και άλλες μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να υπάρχει ένα καλό δικαστικό σύστημα με τη μεταρρύθμιση αυτή. Είναι ένα σύστημα που προστατεύει τους ασθενείς απέναντι στους δυνατούς. Επίσης, ε, το δικαστικό σύστημα δεν θα πρέπει να είναι, να είναι εργαλείο της ε, ανα στιγμή πολιτικής πλειοψηφίας. Όχι. Το δικαστικό σύστημα δεν ενισχύει την κυβέρνηση, ελέγχει την κυβέρνηση. Στη δική μου χώρα, έχουμε τις ε, αποφάσεις στο διοικητικό δικαστήριο που κατά 70% αποφασίζονται υπέρ του πολίτη και όχι υπέρ του κράτους. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτόν τον ορισμό της δικαιοσύνης και να τον εφαρμόσουμε στην πράξη. Θα πρέπει το δικαστικό σύστημα να είναι ανεξάρτητο, να μην ακολουθεί οδηγίες από κάποιους. Επίσης σημαντικό είναι αυτό να λειτουργεί και σε τοπικό επίπεδο. Στην ε, Ανατολική Γερμανία είδαμε μια παρόμοια διαδικασία και τότε μάθαμε ότι πιο σημαντικό για ένα κράτος για να λειτουργεί σωστά είναι τα τοπικά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια. Εκεί έχει επαφή ο πολίτης με το κράτος και γι' αυτό δεν έχει νόημα ε, οι μεταρρυθμίσεις ε, να γίνουν ε, σε ανώτατο επίπεδο μόνο, θα πρέπει να γίνουν από τη βάση. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να προσανατολιστούμε. Θα πρέπει οι πολίτες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στο δικαστικό σύστημα, στο κράτος. Και θα πρέπει ο οικονομικά ασθενέστερος ή μικρομεσαία επιχειρήτηση να προστατευτεί απέναντι στον πιο ισχυρό που έχει στα χέρια του τα εργαλεία της διαφθοράς. Αυτό δεν είναι μόνο κάτι που ρυθμίζει τη συνύπαρξη εντός ενός κράτους, είναι κάτι που σχετίζεται στενά και με τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες ε, για ε, την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά ε, θα ε, προσελκυστούν μόνο εφόσον υπάρχει ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα. Μπορεί κάποιοι να έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά για να έχουμε πραγματικές αποτελεσματικές επενδύσεις χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα, διότι ποιος θα επενδύσει σε μία χώρα που γνωρίζει ότι δεν θα μπορέσει να βρει το δίκιο του. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για το δικαστικό σύστημα μιλάμε έμεσα ή άμεσα και για την οικονομική επιτυχία της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι και βλέπω εδώ τον ε, παλιό μου φίλο Ιωσέγκο που γνωρίζει γιατί μιλάω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you very much. And now... Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Υπουργό Πετρένκο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σόμποντα. που μας δώσατε αυτή ε, τη δυνατότητα να είμαστε εδώ για να σας μιλήσουμε για την πιο σημαντική ε, μεταρρύθμιση στην Ουκρανία. Τα τελευταία 25 χρόνια η Ουκρανία ασχολείται με τις μεταρρυθμίσεις. Όλοι οι προηγούμενοι ε, πρόεδροι, κοινοβούλια είχαν έναν και μόνο στόχο. Ήθελαν να επηρεάσουν το ε, δικαστικό σύστημα και να ελέγχουν τους δικαστές. Αυτό ήταν το πρώτο και κύριο πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν βεβαίως ότι το σύστημα στη διάρκεια των 25 χρόνων μετατράπηκε σε μια πολύ κλειστή δομή, αδιαφανή, διεφθαρμένη, που επέλεγε τους δικαστές, που μόνο κατ' όνομα ήταν δικαστές. Το μεγαλύτερο θέμα ήταν ότι οι δικαστές ήταν το μέσο για την καταπίεση των Ουκρανών πολιτών. Έστελναν τους ανθρώπους στις φυλακές, ε, ε, οι δικαστές εξαρτώνταν τελείων από τους συγγελείς και από τον Γιαννουκόβιτς. Αλλά φτάσαμε σε, ένα, ε, μια φάση που ο ουκρανικός λαός δεν θέλει πια τέτοιο σύστημα. Να σου δώσω, δώσω και άλλη μια στατιστική, ότι το επίπεδο επιβολής των ε, δικαστών έφτανε και το 35% ακόμα και όταν ο πολίτης ελάμβανε την απόφαση ε, στα χέρια του δεν πίστευε την, την απόφαση και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μου τα τελευταία δύο χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω όλου όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή τη μεταρρύθμιση, όλοι οι πυρογνώμονε, οι ΜΚΟ, οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι από όλου του κλάδου, από το Κοινοβούλιο, τη Διεύθυνση τη Προεδρία, ε, γιατί έτσι καταφέραμε την πιο σημαντική μεταρρύθμιση στην Ουκρανία μετά από την ανεξαρτησία μα. Γιατί η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και το να περάσει αυτή η μεταρρύθμιση από το Κοινοβούλιο είναι ένα σπουδαίο μήνυμα για το λαό μας. Η μεταρρύθμιση αυτή δεν έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα της ευρωπαϊκής χώρες. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι για τον λαό μας, τον Ουκρανικό λαό που μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να ε, πιστεύει στη δικαιοσύνη του, να ξέρει ότι θα προστατευθούν τα δικαιώματά του και τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα μέχρι πριν από πέντε χρόνια την φάση του Γιαννουκόβιτς. Γι' αυτό και ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, κατέβηκε στους δρόμους για να απαιτήσει προστασία και κράτος δικαίου. Είμαστε βέβαια στην αρχή ενός ε, πολύ μεγάλου, μιας δύσκολης πορείας, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί και όλα αυτή η νομοθεσία που πέρασε. Πρέπει να σας πω ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος ε, εδώ ανέλαβε ηγετικό ρόλο και το Ουκρανικό Κοινοβούλιο προέβη σε αυτή την ε, αλλαγή του συντάγματος, πρώτη στην ιστορία της Ουκρανίας, είναι η πρώτη αλλαγή του συντάγματος, που το Κοινοβούλιο δηλαδή προβαίνει σε τόσο ριζική μεταρρύθμιση ε, ώστε να αλλάξει και το Σύνταγμα. Πολλοί κόσμος δεν συμπαθεί αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Οι παλιοί δικαστές δεν θέλουν αλλαγές, δεν θέλουν να χαλάσουν τη ζαχαρένια τους και να αλλάξουν το στυλ ζωής τους. Πιστεύουν ότι είναι τιμωρία για εκείνους. Τους εμείς εξηγήσαμε ότι είναι μια ευκαιρία για όλους τους να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, να ανανεωθεί το σύστημα. Και τώρα είναι η ευκαιρία για τη χώρα μας. Γιατί μαζί με την αλλαγή του συντάγματος, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ψήφισε και την εφαρμοστική νομοθεσία γιατί το Σύνταγμα είναι οι βασικές αρχές. Είναι πολύ σημαντικό όμως στην πράξη πώς γίνεται η μεταρρύθμιση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πότε ξεκινάει η μεταρρύθμιση και πότε πρέπει να τελειώσει. Και αυτή η βαρμοστική νομοθεσία δίνει τις απαντήσεις. Ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε την μεταρρύθμιση, ξέρουμε πώς πρέπει να αλλάξει το δικαστικό μας σύστημα, ποιες είναι οι θέσεις για τους νέους δικαστές, ποιες είναι οι αρχές της ανεξαρτησίας τους, και ξέρουμε ακριβώς πότε πρέπει να ολοκληρωθεί και όλα η μεταρρύθμιση. Ο λαός λοιπόν ξέρει ότι μπορεί να έχει το νέο πρόσωπο, το νέο ε, Ουκρανό δικαστή που θα προστατέψει την ελευθερία του που θα ε, ε, προστατεύσει το κράτος δικαίου δεν θα εξυπηρετήσει ούτε το κοινοβούλιο, τον πρόεδρο, το οποιοδήποτε υπάλληλο θα υποστηρίξει και θα προστατεύσει μόνο την Ουκρανική νομοθεσία δεν είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία, είναι πολύ δύσκολη η μεταρρύθμιση και γι' αυτό είναι σημαντική η δική σας υποστήριξη. Η στήριξη από τους φίλους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ σημαντική, διότι δεν έχουμε περιθώριο για λάθη. Και τώρα θα ξεκινήσουν οι πρώτοι διαγωνισμοί για το νότατο δικαστήριο της Ουκρανίας αυτή τη δικασία θα πρέπει να είναι ένα εθνικό ε, σχέδιο. Πρέπει να ζητήσουμε από όλους τους Ουκρανούς ε, νομικούς να έρθουν, να συμμετάσχουν σε αυτούς τους ε, διαγωνισμούς, ώστε να γεμίσουν με νέους ποιοτικούς δικαστές τα Ουκρανικά δικαστήρια. Πρέπει αυτό να ολοκληρωθεί μέσα στου επόμενου έξι μήνε. Να είναι ένα πρώτο μήνυμα ότι το Ουκρανικό δικαστικό σύστημα θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη του Ουκρανικού λαού και τη Ουκρανική κοινωνία. Μετά έχουμε μια άλλη σειρά διαγωνισμών για ε, να επανδρωθούν τα τοπικά ε, δικαστήρια και πρωτοδικεία αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό να επιτύχουμε το ανώτατο δικαστήριο με 200 νέους δικαστές που θα περάσουν δημόσιους διαγωνισμούς διαφανείς, θα περάσουν έλεγχο κατά, ε, ε, κατά τη διαφθοράς και οι Ουκρανοί πολίτες θα δουν όλους αυτούς τους υποψήφιους και θα καταλάβουν ότι θα μπορούν να έχουν και πάλι εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου those people who have dignity and honor. Ότι επανήλθαν οι αξιοπρεπείς και έντιμοι άνθρωποι στα δικαστήρια. Χρειαζόμαστε πραγματικά την υποστήριξη των τεχνικών ομάδων για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους διαγωνισμούς, να είναι διαφανείς οι συνθήκες, να παρακολουθήσουμε και να ελέγξουμε τους υποψηφίους και μετά να διδάξουμε σε αυτούς τους νέους δικαστές που θα αποτελούν το νέο δικαστικό σύστημα στην Ουκρανία και θα ήταν πολύ καλό να μπορέσουμε αυτό να το συζητήσουμε σήμερα. Είμαστε ανοιχτοί να δώσουμε όλες τις απαντήσεις και όλες τις λεπτομέρειες για αυτή τη μεταρρύθμιση. Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε όλες τις συστάσεις. Κανένας δεν, μπορεί να πει ότι η Ουκρανία κάνει ριζική αλλαγή στο δικαστικό τομέα και ότι η, η μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών είδαμε να ανοίγεται μια ευκαιρία, ένα παράθυρο, μια ευκαιρία για ανανέωση και του προσωπικού των δικαστηρίων και του δικαστικού συστήματος και αυτό να γίνει με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο σημαντικό θέμα της μεταρρύθμισης είναι και η μεταρρύθμιση του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. καθώς και η μεταρρύθμιση του συστήματος δικαστικής αρρωγής. Γιατί το κράτος πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε όλους και στους φτωχότερους των φτωχών να έχουν νομική βοήθεια. Η πιο σημαντική μεταρρύθμιση είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντικό να επιτύχει και το Κοινοβούλιο σας έλαβε ιστορική σημασία σε απόφαση. Όπως και το δικό μας που πέρασε αυτή τη μεταρρύθμιση και τώρα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να η κυβέρνηση, η ΜΚΟ και ο δημόσιος τομέας να εφαρμόσουμε τη μεταρρύθμιση και να θεσπίσουμε ένα πραγματικά ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα που θα προστατεύει όλους τους Ουκρανούς. We don't have another Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στο λαό μας που έκανε την επανάστασή του. Η επιτυχία μας θα σημάνει ότι η Ουκρανία έχει αλλάξει και όλες οι άλλες μεταρρυθμίσεις και σε τους υπόλοιπους τομείς θα είναι επιτυχής εάν καταφέρουμε σωστά τη μεταρρύθμιση της ε, δικαιοσύνης. έτσι ώστε ο κόσμος ε, και οι περιοδητές στην Ουκρανία, αν ξέρουν ότι θα μπορούν να έρθουν ε, στην Ουκρανία και θα μπορούν να στραφούν στη δικαιοσύνη και να βρουν το δίκαιο τους, θα έρθουν περισσότεροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Και νομίζω τώρα θα πρέπει να αλλάξουμε θέσεις για να δώσουμε τη θέση μας ε, στους ομιλητές του πρώτου πάνελ, της πρώτης συζήτησης. Τον κύριο Φιλάτοφ, την κυρία το τον κύριο Βριάντ, τον κύριο Κοζιακόφ και τον κύριο Κούμπιντα. Ελάτε παρακαλώ. Uh, αγαπητοί συναδέλφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ξεκινάμε τώρα την πρώτη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος και του συντάγματος, συγγνώμη, του δικαστικού συστήματος. Δίνω το λόγο στην κυρία Οξάνα Σιρόιντ, αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου του Φερκόβνα Ράντα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Μια μεγάλη ευκαιρία το να βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να συζητήσουμε αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία. Ζητήματα που απαιτούν κατανόηση και συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε. Ξεκινώντας, θα αναφερθώ στα πρόσφατα γεγονότα για ε, την εξυγίανση του δικαστικού συστήματος που αναφέρθηκε ε, και από τους προηγούμενους ομιλητές. Είδα ότι υπάρχει ελπίδα ελπίδα μεταξύ της κοινή γνώμης ότι αυτή τη φορά το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και διαφορετικό. είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της μεταρρύθμισης και κατά τη συνέντευξη τύπου που έγινε λίγο νωρίτερα, όταν τα λέγαμε αυτά, όπου είδα την ίδια ελπίδα στα μάτια των ακροατών της συνέντευξη τύπου, είδα ότι για τη μεταρρύθμιση του συντάγματος και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμη. Και δεν γίνονται εν μια νυχτή όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε. Και ελπίζουμε ότι Έφτασε αυτή η στιγμή της αφετηρίας όταν ψηφίστηκαν οι τροποποιήσεις του συντάγματος. Χρειάζονται για τη μεταρρύθμιση τουλάχιστον δύο παράμετροι. Πρώτον, καλή νομοθεσία και δεύτερον, εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη και πίστη στην υλοποίηση του νέου νόμου και για το Σύνταγμα και για την εφαρμοστική νομοθεσία ε, ε, θεωρώ ότι είναι σωστά νομικά κείμενα, των οποίων η υλοποίηση μπορεί να γίνει σωστά προς όφελος των πολιτών της Ουκρανίας. Όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει όλοι να καταβάλουμε από κοινού προσπάθειες και να είμαστε αποφασισμένοι και επί χρόνια, επί δεκαετίες θα έλεγα μπορεί να χρειαστεί αυτό, να συνεργαστούμε και να προσπαθούμε γιατί μπορεί να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορεί να μην είναι η δική μας γενιά πολιτικών ε, που ε, θα ολοκληρώσουν αυτή την προσπάθεια, αλλά και άλλοι μετά από εμά θα συνεχίσουν. Μιλώντας ε, για την νομοθεσία, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτές οι τροποποιήσεις του συντάγματος και ε, αυτή είναι η νόμη είναι πολύ σημαντική. Αλλά δεν ολοκληρώθηκε το έργο μας. Υπάρχει ακόμη ένας μακρύς κατάλογος τροπολογιών που πρέπει να εγκριθούν για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. χρειάζεται νομοθεσία για το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών, γιατί αυτός είναι ο θεσμός που έχει το βασικό ρόλο για την επιλογή και για τα πειθαρχικά ζητήματα των δικαστών. Τροπολογίες των δικονομικών κωδίκων έχοντας πάντοτε κατά νου ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την έννοια της ε, δικαιοσύνης που τα τελευταία χρόνια έχει υπονομευθεί. Και επίσης πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η μεταρρύθμιση του ποινικού συστήματος της ποινική δικαιοσύνης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πρέπει και αυτό να το προωθήσουμε. Και όταν μιλάμε για τον ε, τομέα του ποινικού δικαίου, πρέπει να τονίζουμε ιδιαίτερα τη δημιουργία ενός δικαστηρίου κατά της διαφοράς. Και στο νόμο για το καθεστώς των δικαστών αναφέρεται αυτό, αλλά χρειάζεται ε, πολλή δουλειά να γίνει και αναμένω και μεγάλη υποστήριξη από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα δικαστήριο κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στο κράτος. Θα πρέπει όλες οι υποθέσεις διαφθοράς να εξεταστούν με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο και το βασικότερο είναι να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των ανθρώπων που θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Και εδώ θα χρειαστούμε και τη δική σας βοήθεια. Μιλώντας για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι που δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς ε, την ε, ολοκληρωτική μεταρρύθμιση του συστήματος ε, των νομικών των δικηγόρων που εκπροσωπούν στο δικαστήριο. Χρειάζεται ένα αυστηρό σύστημα επιλογής και πειθαρχικό σύστημα παράλληλα. Χαίρομαι που είναι εδώ και ο Γενικός Εισαγγελέας, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα χωρίς να γίνει μεταρρύθμιση και ε, της εισαγγελίας. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη λειτουργία και το ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα και του γραφείου του ή της Γενικού Εισαγγελέως και να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του εισαγγελέα καθώς και το τι θα λογοδοτούν. Τελευταίο και όχι έσχατο είναι η μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης των δικαστών. Η μεγάλη διαφθορά στα δικαστήρια συχνά ξεκινάει από τα πανεπιστήμια, από τη διαφθορά που υπάρχει στη νομική εκπαίδευση. Και δεν είναι και μεγάλο μυστικό στην Ουκρανία ότι σε όλους αυτούς τους τομείς επικρατεί διαφθορά. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα και στο σύστημα της παιδείας και της εκπαίδευσης των νομικών και ως, το, προς το περιεχόμενο και ως προς τη μέθοδο εκπαίδευσης, γιατί στην Ουκρανία συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τη σοβιετική μέθοδο εκπαίδευσης. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς εσάς, διότι εσείς έχετε τη γνώση και την εμπειρία, καθώς και την νομιμοποίηση που μπορεί να μας βοηθήσει να το κάνουμε. Καλόπιστη υλοποίηση λοιπόν είναι αυτό που θέλουμε μέσα σε τρεις μήνες θα αντιμετωπίσουμε την πρώτη πρόκληση που θα είναι και δοκιμασία για το αν μπορούμε να το κάνουμε. Επιλογή των δικαστών του Ανωτάτου Συμβουλίου, δεύτερον πειθαρχικό σύστημα και αποπομπή όλων των διεφθαρμένων δικαστών, τρίτον δίωξη και λογοδοσία για τους διεθερμένους ιδίως δικαστές αλλά και εισαγγελείς, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν υλοποιούμε κάτι, γιατί μπορούμε να εφαρμόζουμε κανόνες που μπορούν να αποβούν σε καλό ή σε κακό, όπως παραδείγματος χάρη το μονοπόλιο των δικαστηρίων. Η κοινωνία των πολιτών ανησυχεί και πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε συγκεκριμένους κανόνες στην πράξη. Βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε περιλαμβάνουν την παρουσία της Ρωσίας και δεν μιλώ για τη στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία. Πρέπει να κατανοήσετε ότι η Ρωσία υποστηρίζει και υποστήριζε δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι θα αντιδράσουν και θα αντισταθούν πάρα πολύ σε αυτή τη μεταρρύθμιση διότι θέλουν να αποτύχει κάθε μεταρρύθμιση στην Ουκρανία και αυτή η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ακόμη περισσότερο. Άλλη πρόκληση για μας είναι ο τομέας της εμπιστοσύνης. Πιστεύω και εδώ ότι η συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Θυμάμαι ένα παράδειγμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όταν είχαμε έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είδαμε τη διαφορετική κουλτούρα επικοινωνίας. Είναι πολύ ευάλωτη ακόμη αυτή η κουλτούρα της επικοινωνίας στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο, αλλά είναι κάτι για το οποίο αποτέλεσε ένα πόλο διαφωτισμού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακόμη θυμάμαι από προσωπική εμπειρία όταν ψηφίσαμε τις τροπολογίες του συντάγματος την πρώτη φορά ε, μίλησα με τους κύριους συνομιλητές μου που όλοι βρίσκονται εδώ σε αυτήν την αίθουσα σήμερα και είπαμε ότι στη δεύτερη ψηφοφορία θα χρειαστούμε και την εφαρμοστική νομοθεσία. Επί προσπαθούσαν να συνεργαστούν όλοι οι αρμόδιοι με τους φόβους τους, ε, προσπαθώντας να χτίσουν την εμπιστοσύνη τους και έτσι καταλήξαμε στο να ψηφιστούν οι νόμοι. Το θέμα της εμπιστοσύνης αναφέρθηκε ήδη πολλές φορές και σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό για να έχουμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο προηγούμενος ομιλητής μίλησε για νέα νοοτροπία και νέες σχέσεις και νομίζω ότι στο όνομα όλων των ε, μελών που είναι παρόντα Μία από τις ε, πιο συγκινητικές ε, στιγμές ε, ήταν η υπογραφή της συμφωνίας. Πράγματι, λοιπόν, υπάρχει πολύ στενή σχέση. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και δίνω το λόγο στον κύριο Λέξη Φιλατόφ, αναπληρωματικό διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου. Δέκα λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω εδώ σήμερα και να συζητήσουμε το πολύ σημαντικό θέμα της δικαστικής μεταρρύθμισης της Ουκρανίας. Μάλλον δεν θα μιλήσω για τη σημασία της μεταρρύθμισης του δικαστικού. Οι προλαλήσαντες νομίζω το συζήτησαν αρκετά. Δεν νομίζω ότι είναι επίμαχε θέμα, αλλά το δικαστικό σύστημα της Ουκρανίας έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα προβλήματα δεν είναι μόνο η διαφθορά. Δεν είναι μόνο το χαμηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Δεν είναι η ανεξαρτησία. Εάν όμως πάρουμε όλα τα προβλήματα μαζί και δούμε το επίπεδο εμπιστοσύνης των Ουκρανών στο δικαστικό, στο δικαστικό τους σύστημα, θα εκπλαγείτε. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να πούμε ότι και η εμπιστοσύνη απέναντι στο Κοινοβούλιο ή την κυβέρνηση δεν είναι πολύ ψηλό. Αλλά όταν ο κόσμος δεν εμπιστεύεται το δικαστικό σύστημα, αυτό δείχνει σημαντικά προβλήματα στην κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε δικαστής είναι διαφθαρμένος ή ότι κάθε απόφαση λαμβάνεται με μη επαγγελματικό τρόπο. Αλλά τα προβλήματα αυτά απαντώνται πολύ συχνά και μάλιστα πολύ πιο συχνά από ό,τι θα περίμενε κανείς σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Γνωρίζετε ότι μία από τις προτεραιότητες του Προέδρου στην στρατηγική του 2020 ε, ήταν η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Πριν σχεδόν δύο χρόνια, ο Πρόεδρος ε, δημιούργησε ε, έναν ανεξάρτητο φορέα, το, την Επιτροπή για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, όπου συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς για να εκπονήσουν ένα σχέδιο δράσης ώστε να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι αποτελέσματα πρέπει να πετύχουμε στην μεταρρυθμίση αυτή. Οι στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν Ήταν μεταξύ άλλων ε, μια ισχυρή δικαιοσύνη, ανεξάρτητη. Ε, θα σας δείξω και τις διαφάνειες. Ε, δεν είμαι βέβαιος ότι φαίνονται ολόκληρες οι διαφάνειες, αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειαζόμαστε λοιπόν υψηλά επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα ε, για τον δικηγορικό σύλλογο. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική εισαγγελία, νέο σύστημα εφαρμογή ε, των δικαστικών αποφάσεων, ε, διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για παράδειγμα, επικρίνει όχι τόσο πολύ την ποιότητα των δικαστηρίων και των ε, δικαστικών αποφάσεων, αλλά στο χαμηλό ποσοστό εφαρμογής ε, των αποφάσεων. Και επίσης χρειαζόμαστε βελτιωμένο, ε, βελτιωμένη νομική κουλτούρα. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι πολύπλοκο. Δεν αρκεί να τροποποιήσουμε την ομοθεσία και έτσι την επόμενη μέρα ή τον επόμενο μήνα να έχουμε ξαφνικά κράτος δικαίου στη χώρα. Είναι κάτι που σχετίζεται και με τους θεσμούς και ακόμα περισσότερο σχετίζεται με τους ανθρώπους. Η νομοθεσία είναι μεν ατελής, όχι όμως στο βαθμό που προκαλεί όλα τα προβλήματα στο δικαστικό σύστημα της Ουκρανίας. Πρέπει να γίνουν πολλά για τροποποίηση της νομοθεσίας, αλλά το πιο σημαντικό μέρος της μεταρρύθμισης ε, είναι να ασχοληθούμε τους ανθρώπους αυτούς, όχι μόνο τους δικαστές, αλλά και τους ε, εισαγγελείς, τους δικηγόρους κλπ. και γι' αυτό έχουμε εντοπίσει κάποια στοιχεία της μεταρρύθμισης. Ε, καταρχάς, ε, τροποποίηση της ε, νομοθεσίας. Το Σύνταγμα αποτελεί τη βάση για ένα νέο ποιοτικό σύστημα. Επίσης, χρειαζόμαστε κάποιες κανονιστικές τροποποίησεις το δικαστικό σύστημα, το καθεστώς των βουλευτών, νέος κανονισμός των δικαστηρίων, ο νέος νόμος για το δικηγορικό σύλλογο και η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων όσον αφορά τους ε, θεσμούς ε, θα πρέπει ε, να έχουμε επανεκκίνηση κάποιων φορέων όπως είναι το υψηλό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε με την αξιολόγηση των βουλευτών. Και αυτό σχετίζεται με αυτό που σας είπα πριν, το ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους. Ποια είναι λοιπόν η πρόοδος που έχει σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2015 το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας υιοθέτησε τον ε, νόμο για την ε, δίκαιη δίκη που έλυνε μια σειρά πρακτικών προβλημάτων ε, που μπορούσαν να λυθούν χωρίς τροποποίηση του συντάγματος. Ο νόμος αυτός έχετε επιτρέψει ανανέωση της ε, λειτουργίας ε, της ε, Υψηλής Επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαστών σύμφωνα με τους νέους διαφανείς κανόνες. Το επόμενο βήμα ήταν τροποποίηση του συντάγματος. Και η αρμόδια επιτροπή που συγκλήθηκε πέρσι τον Απρίλιο έχει συνεργαστεί στενά με την ε, Επιτροπή για το Δικαστικό Σύστημα και έχει, υποσ... έχει λάβει πολλή υποστήριξη. Ε, για παράδειγμα, ήταν ιδιαίτερα ποιοτικό το σχέδιο κειμένου που έλαβε. Ο νόμος για τροποποίηση του συντάγματος υιοθετήθηκε πρόσφατα στις 2 ε, Ιουνίου φέτος και υιοθετήθηκε μαζί με το νέο νόμο για το δικαστικό σύστημα και το καθεστώς των βουλευτών, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Επίσης ε, έχει ασχοληθεί με το θέμα της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων και έχουμε δύο νέους νόμους για τις διαδικασίες εκτέλεσης ε, των δικαστικών αποφάσεων ε, καθώς και τις λειτουργίες των υπαλλήλων των δικαστικών λειτουργών κλπ. Και επίσης έχουμε και νέο νόμο για το δικηγορικό σύλλογο. Οι λύσεις κλειδιά που έχουν εισαχθεί με αυτές τις νομοθετικές τροποποιήσεις ε, συμπεριλαμβάνουν από πολιτικοποίηση και ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος. Ε, δικαστήρια μπορούν να δημιουργηθούν ή να διαλυθούν μόνο με νόμο. Επίσης, ε, έχουν ε, απομακρυνθεί όλοι οι πολιτικοί φορείς από την ε, διαδικασία διορισμού των δικαστών και επίσης υπάρχει πολιτική ουδετερότητα των μελών του Υψηλού Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με δημιουργία αποτελεσματικού και υπεύθυνου συστηματικού συστήματος, όχι μόνο εξάρτητου δηλαδή. Υψηλότερα πρότυπα για του δικαστές, περιορισμό της ασυλίας τους και πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για απόλυση τους. Επίσης, εγγυήσεις ε, κατά της διαφθοράς, για παράδειγμα, Ε, λόγοι που σχετίζονται με το εισόδημα του δικαστή που μπορούν να οδηγήσουν στην απόλυσή του. Κατόπιν έχουμε επανεκκίνηση του δικαστικού συστήματος, ε, έχουμε τις ε, ατομικές αξιολογήσεις, μια ειδική διαδικασία που έχει εισαχθεί και σχετίζεται με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Αυτή η ειδική αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια επαγγελματικής ε, ε, ικανότητας, σε συνηθική και ακαιρεότητα του δικαστή. Κάθε δικαστής περνάει από τη διαδικασία αυτή για να ε, επιβεβαιώσει ότι συμμορφώνεται με τα κριτήρια αυτά. Οι νέοι δικαστές θα προσλαμβάνονται με βάση διαγωνισμούς και επίσης ε, προβλέπεται ε, συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών, κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν. Και βέβαια μια από τις πιο σημαντικές λύσεις που σας ανέφερα ήδη επανειλημμένα είναι η δημιουργία του νέου ανώτατου δικαστηρίου. Ουσιαστικά από το μηδέν. Η τροποποίηση του συντάγματος ε, συμπεριλαμβάνει και εισαγωγή ευρωπαϊκών προτύπων για την ε, οργάνωση και λειτουργία της εισαγγελίας ε, καθώς και ενίσχυση του δικηγορικού συλλόγου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε ένα καλό και υψηλής ποιότητας δικαστικό σύστημα. Λίγα λόγια σχετικά με την αξιολόγηση των δικαστών. Ξεκίνησε φέτος τον Φεβρουάριο η διαδικασία για την αξιολόγηση των βουλευτών. Ακόμα και για πολλούς ικανονούς ήταν αναπάντεχα τα αποτελέσματα. Πάνω από 300 δικαστές πέρασαν τη διαδικασία αξιολόγησης και περίπου το 40% δεν πέρασαν επιτυχώς την αξιολόγηση. Κάτι που δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο δικαστικό τομέα. Μας περιμένει όμως πολλή δουλειά ακόμα. Το 2016 περιμένουμε νέους ε, κανόνες ε, για τη λειτουργία των δικαστηρίων και το νέο νόμο για τον Δικηγορικό Σύλλογο και περιμένουμε επίσης νέα νομοθεσία για τη νομική εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Σέγγι Κοζιάκοφ ε, πρόεδρο της ε, Επιτροπής Αξιολόγησης. Για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω αυτήν την εισήγηση. Η η Επιτροπή Εξολόγησης Προσόντων των Δικαστών είναι ένα μόνιμο σώμα στο δικαστικό σύστημα της Ουκρανίας. Όλα τα προηγούμενα μέλη αυτής της Επιτροπής απολύθηκαν τον Απρίλιο του 2004 μέσω της νομοθεσίας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο δικαστικό σύστημα της Ουκρανίας. Το Δεκέμβριο του 2014, μετά από 9 μήνες διάλειμμα, η Επιτροπή άρχισε να εργάζεται για τη νέα σύσταση. Τώρα αποτελείται από 14 μέλη, 10 εκ των οποίων είναι δικαστές ή συνταξιούχοι δικαστές και τέσσερις είναι ε, νομικοί και καθηγητές δικαίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι πανεπιστημιακός καθηγητής και πρώην εισαγγελέας. Η νομοθεσία επιτρέπει σε αυτή την Επιτροπή, ε, δίνει μάλλον διάφορες αρμοδιότητες όσον αφορά το τομέα της δικαστικής σταδιοδρομίας. Ε, αυτές είναι η επιλογή των υποψηφίων για την θέση ε, δικαστή, η έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών όσον αφορά τους δικαστές τοπικών και τοπικών δικαστηρίων και εφετείων, η μεταφορά ενός δικαστής σε άλλα δικαστήρια και ε, ε, ούτω καθεξής. Η νέα νομοθεσία αφορά την εφαρμογή όλων, όλες τις νέες διαδικασίες που αφορούν αυτήν τη νέα νομοθεσία η δε δεξιότητες, μάλλον αξιολόγηση των προσόντων των δικαστών αποτελεί τη πιο σημαντική ε, εργασία αυτής της Επιτροπής. Όλοι οι δικαστές πρέπει να περάσουν από την αξιολόγηση. Υπάρχουν περίπου 8.000 δικαστές στη χώρα και η Επιτροπή μας πρέπει να κάνει αξιολόγηση για όλους. Δεν υπάρχει προηγούμενο για κάτι τέτοιο στην ευρωπαϊκή πρακτική, είναι αλήθεια. Ωστόσο, η ε, διαδικασία αξιολόγησης εγκρίθηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η ανάπτυξη και η έγκριση όλων των εγγράφων εντός της αξιολόγησης έγινε από την Επιτροπή με την ε, στήριξη εμπειρογνωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και κατέστη πραγματικά και εναλλακτική λύση για την απαλλαγή από τους παλιούς δικαστές, πράγμα που ζήτησαν όλοι οι πολιτικοί αλλά και ο ουκρανικός λαός. Η αξιολόγηση αποτελείται από τέσσερα στάδια. Πρώτον, έχουμε μια ανώνυμη εξέταση από έναν δικαστή και έπειτα επαλήθευση του φακέλου του δικαστή και συνέντευξη. Οι αρχικές ε, η αρχική μάλλον αξιολόγηση των δικαστών που αναφέρθηκε από το συναδέλφο σήμερα ξεκίνησε το, ε, το Φεβρουάριο του 2016 στη διάρκεια τεσσάρων μηνών η Επιτροπή έκανε την πρώτη αξιολόγηση ε, σε σχέση με περίπου 400 ε, δικαστές. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά όχι μόνο για την Επιτροπή μας αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία και όπως αναφέρθηκε το 40% των δικαστών δεν ακολούθησαν αυτή τη διαδικασία, αλλά περίπου 60% των δικαστών αντιμετώπισαν ε, το θέμα της προσαρμογής στα τοπικά δικαστήρια. Μάλιστα, 30% ε, των δικαστών ε, παρετήθηκαν πριν αρχίσει η διαδικασία εξολόγησης ή δεν προσήλθαν ε, γιατί φοβούνται απλώς να μιλήσουν με τα μέλη της Επιτροπής για τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί από την Εθνική Υπηρεσία ε, καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης, ε, διάφοροι ζήτησαν διαλύματα για να μπορέσουν να επαληθεύσουν το νομικό φάκελο Ιδιαίτερα όσον αφορά το γραφείο, την, την υπηρεσία μάλλον καταπολέμησης της διαφθοράς και γι' αυτό και έτσι ξεκίνησε η επαλήθευση της ε, του δικαστικού ε, συστήματος. Άλλες ε, διαδικασίες έδειξαν ότι Ε, ε, θα έπρεπε να έχουν καλύτερη γνώση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τους όσους πέρασαν την αξιολόγηση το χειμώνα ή τις αρχές της Άνοιξης. Άρχισαν να μαθαίνουν και να εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατέστησαν πιο υπεύθυνοι απέναντι στις αποφάσεις που λαμβάνονταν από τα το ανώτατο δικαστήριο, οι δικαστές έδειξαν ότι δεν ότι εκτιμούν την κατάσταση, δεν έρχονται με, αυτή, με ακριβά αυτοκίνητα, ούτε ντυμένοι με ακριβά ρούχα και ρολόγια κατάλαβαν ότι η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Διαφθοράς γνωρίζει τους κινδύνους διαφθοράς όσον αφορά τα πάνες που ξεπερνούν το εισόδημα ενός δικαστή. Στις 6 Ιουνίου φέτος υιοθετήθηκε η μεταρρύθμιση της, ε, του δικαστικού σώματος από το, από το Κοινοβούλιο μας και το νέο καταστατικό για τους δικαστές. Έχουμε νέα κριτήρια για την αξιολόγηση των δικαστών και εκεί εντάσσεται και η λέξη ακαιρεότητα. Να αναφέρω ακόμα μια φορά πως είναι υποχρέωση της Επιτροπής μας να προσφέρει μια νέα ανταγωνιστική ε, πρόταση για την επιλογή των νέων ε, δικαστών για το Ανώτατο Δικαστήριο. Μέχρι 200 δικηγόροι θα εκλεγούν στο Ανώτατο Δικαστήριο ε, σε διαφανή βάση για να είναι κανείς υποψήφιος για τη θέση δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ουκρανίας. Ε, ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να έχει εργαστεί ως εισαγγελέας για μίνιμουμ 10 χρόνια. Ε, αναζητούμε ουσιαστική βοήθεια από την υπηρεσία κατά της διαφθοράς καθώς και το γραφείο ε, κατά της διαφθοράς για να αναλύσουμε πιθανούς κινδύνους διαφθοράς για τους υποψήφιους ε, σε δικαστικά αξιώματα. αναμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία επιλογής μέσα στο 2016 και έτσι να έχουμε έναν καθοριστικό αντίκτυπο στο δικαστικό σύστημα της Ουκρανίας για τα επόμενα χρόνια. Επίσης με χαρά μπορώ να σας ενημερώσω ότι έχουμε προετοιμάσει ένα βίντεο για τη διαδικασία Αξιολόγηση των προσόντων, όπου δικαστές με διαφορετικά επίπεδα ε, ε, προσόντων ε, παρουσιάστηκαν και με την άδειά σας θα ήθελα να σας δείξουμε αυτό, αυτή την ταινία μάλλον να σας την στείλουμε και μπορείτε να την προωθήσετε και στους ενδιαφερόμενους βουλευτές. Να τονίσω ότι είναι η πρώτη φορά που η μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος γίνεται υπό καθεστώς ε, στρατιωτικής ε, κατοχής ενός τμήματος της επικράτειάς μας. Ωστόσο, πρόκειται για μια επιτυχή διαδικασία ε, που δείχνει πόσο δυναμική και είναι αυτή η διαδικασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω να δείτε και εσείς τα θετικά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και για τις σημειώσεις που μας δώσατε. Έχουμε τυπώσει κάποια αντίγραφα και μπορούμε να τα μοιράσουμε σε όποιον επιθυμεί να έχει ένα αντίτυπο. Και τώρα θα δώσω λόγο στον Ειδικό Σύμβουλο για την Ουκρανία, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δέκα λεπτά και πάλι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σβόμποντα που καλέσατε το Συμβούλιο της Ευρώπης σε αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ουκρανία. Ομιλώ ως πρόσφατα οριστής και εκ μέρους του κυρίου τόρβγιαν Νάγκεντ και Ζητώ συγγνώμη εκ μέρου ε, του κυρίου Χρήστου Γιακουμόπουλου, που ήταν ο προηγούμενο ειδικό σύμβουλο. Ήθελε να συμμετάσχει, αλλά τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η πτήση του και δεν μπόρεσε να φτάσει στις Βρυξέλλες. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει πολύ ενεργό ρόλο στην Ουκρανία και συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά θέματα. Ο τομέας της δικαιοσύνη είναι ένας από τους τομείς, αλλά δεν είναι η μοναδική δραστηριότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης που εκπροσωπείται ευρύτατα στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα γραφείο του Συμβουλίου της Ευρώπης με αρκετού συμβούλους που εργάζονται για διαφορετικά θέματα στην Ουκρανία. Το Συμβουλίο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε ένα σύστημα, ολοκληρωμένο σύστημα δράσεων για την Ουκρανία, οι οποίες διεξάγονται σε συνεργασία με τις Ουκρανικές Αρχές. Το Συμβουλίο της Ευρώπης χαιρετίζει και ο Γενικός Γραμματέας έκανε μια δήλωση χαιρετίζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις, ιδίως τις τροπολογίες του συντάγματος και την νέα νομοθεσία για το δικαστικό τομέα και το καθεστώς των δικαστών. Ο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου τη Ευρώπη θεωρεί πολύ σημαντικά βήματα αυτέ τι νέε εξελίξει και η μεταρρύθμιση αυτή φαίνεται ότι ετοιμάζει το δρόμο για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι βασικοί πυλώνες ε, που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες βάσει του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεσματικό, ε, ανταγωνιστικό και ικανό ε, δικαστικό σώμα χωρίς διαφορά αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση αυτών των αρχών. Θα σας πω δύο λόγια τώρα και για αυτές τις βασικές μεταρρυθμίσεις. Η πρώτη μεταρρύθμιση ήταν η τροπολογία του, οι τροπολογίες του συντάγματος. Οι τροπολογίες αυτές εγκρίθηκαν στις 2 Ιουνίου και ανταποκρίνονται στις περισσότερες συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως της Επιτροπής της Βενετίας για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου. Η Επιτροπή της Βενετίας συνεργάστηκε στενά με την Συνταγματική Επιτροπή του Φερχόμνα Ράντα του Ουκρανικού Κοινοβουλίου και οι περισσότερες συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας αντικατοπτρίζονται στο νέο κείμενο. Ο νόμος για το δικαστικό σώμα και το καθεστώς των δικαστών όταν θα υλοποιηθεί θα εγκαθιδρύσει ένα δικαστικό σύστημα που θα είναι συμβατό με τα πρότυπα και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η μεταρρύθμιση του εισαγγελικού σώματος που ξέρω ότι είναι θέμα της επόμενης συζήτησης, αλλά θέλω να το αναφέρω, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης χαιρετίζει τον διορισμό του κ. Λουτσέγκο ως νέου Γενικού Εισαγγελέα. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης τον έχει ενημερώσει για την υποστήριξη ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης και για την δέσμευσή μας να συνεργαστούμε προς ε, τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, είναι όλες αυτές τις αλλαγές να τις υλοποιήσουμε. Οι αλλαγές ε, των νομοθετικών κειμένων ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να περάσουμε στη δημιουργία ενός νέου δικαστικού τομέα στην Ουκρανία, αλλά χωρίς σωστή υλοποίηση όλες αυτές οι αλλαγές δεν θα έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υλοποίηση είναι μια μακρά οδός που θα απαιτεί δέσμευση και αποφασιστικότητα από όλους τους θεσμικούς φορείς και όλους τους εμπλεκομένους. Το Συμβουλίο της Ευρώπης θα συνεχίζει να υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση και να συνεργάζεται με όλους τους φορείς και όλες τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη μεταρρύθμιση, ώστε να επιτευχθεί ο κοινό μας στόχος. Κυρίες και κύριοι, όλη αυτή η δουλειά που γίνεται αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. Εφόσον η εμπιστοσύνη προς το δικαστικό σώμα και προς το κράτος είναι βασικό, ε, βασική προϋπόθεση για την δημοκρατία στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Και τελευταίος ομιλητής για αυτή την πρώτη συζήτηση θα είναι ο κύριος Ρόμαν Κουίμπιντα από το Κέντρο Πολιτικής και Νομικής Μεταρρύθμισης. Δέκα λεπτά και για σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στη σημερινή εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, συμφωνώ απολύτως με τους προλαλήσαντες ότι οι νόμοι που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες ε, μας έδωσαν μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσουμε και να διεξάγουμε την ε, δικαστική μεταρρύθμιση στην Ουκρανία σύμφωνα με δυτικά πρότυπα. Οι πολίτες ανέφεραν τα εξής τα βασικά προβλήματα του συστήματος. Διαφθορά στους δικαστές, εξάρτηση των δικαστών από ολιγάρχες και πολιτικούς ε, ε, και αμοιβαία συγκάλυψη εντός ε, των δικαστηρίων. Μία έρευνα που έγινε φέτος έδειξε ότι οι περισσότεροι πολίτες γενικά στηρίζουν τα μέτρα που περιγράφονται στις συνταγματικές τροποποιήσεις. Για παράδειγμα, επανεξέταση όλων των δικαστών, απομάκρυνση των πολιτικών φορέων ε, από, τον διορισμό, από τις διαδικασίες διορισμού των ε, δικαστών, ε, περιορισμό των ασυλιών των δικαστών, να μπορεί να γίνει προσωπική προσφυγή κατά των θεσμών κλπ. Θα πρέπει να καταλάβουμε τις βασικές προκλήσεις για μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Ε, δεν μπορώ να σας πω πώς θα ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Σημαντικό όμως είναι να ε, εντοπίσουμε τις προκλήσεις. Καταρχάς, οι περισσότεροι πολίτες ε, δεν πιστεύουν ότι θα πετύχει η δικαστική μεταρρύθμιση που ενέκρινε αυτό το μήνα το Κοινοβούλιο. Αυτό δεν έχει, γίνει, δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας ε, κοινωνιολογικής μελέτης, αλλά συνομιλώ με Ουκρανούς ε, δραστήριους ε, στην κοινωνία των πολιτών και μόνο το 25-30% τους πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει μια τέτοια μεταρρύθμιση. Και ε, οι λόγοι για αυτή τη χαμηλή εμπιστοσύνη επικύλουν. Ε, καταρχάς υπάρχει γενική δυσαρέσκεια και αγανάκτηση με την πολιτική. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό ε, αποτελεί συγκέντρωση εξουσίας από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος ε, μπορεί να αποφασίσει τη δημιουργία ή διάλυση δικαστηρίων, ε, την ε, απόσπαση ή την προαγωγή των δικαστών. Οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των δικαστών και το υψηλό Συμβούλιο Δικαιοσύνης θα μπορέσει να απομακρύνει τους διεφθαρμένους δικαστές από το σώμα των δικαστών δεν εκπροσωπούνται μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, στι δύο ε, επιτροπές αυτές. Έτσι υπάρχει ακόμα ο φόβος για αμοιβαία συγκάλυψη. Ε, μετά έχουμε την αντίσταση από πλευράς ε, των δικαστών. Το συνταγματικό δικαστήριο αναμένεται να λάβει μεγάλη σειρά συνταγματικών προσφυγών. Η τρίτη πρόκλησή μας ε, είναι ότι οι πολιτικοί θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την επιρροή τους ε, στο δικαστικό σύστημα παρά ε, την κατάργηση κάποιων μηχανισμών. Και έτσι θα μπορέσουν οι νέες μέθοδοι να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν οι πολιτικοί δικούς τους δικαστές, ενώ άλλα δικαστήρια θα διατηρήσουν το άτυπο σύστημα επιρροής μέσω των ε, δικαστών τους. Επίσης, το δικαστήριο για την διαφθόρα είναι δικαστήριο πρωτοβάθμιο το καθεστώς αυτού του δικαστηρίου δεν ε, έχει, ε, έχει έγκαια όσον αφορά την ανεξαρτησία του, την ε, επιλογή των δικαστών κλπ οι πολιτικές αρχές φαίνεται να μην έχουν πραγματικά την πρόθεση να δημιουργήσουν ένα τέτοιο δικαστήριο. Οι εμπειρογνώμονες επίσης έχουν, έχουν εντοπίσει άλλα προβλήματα όσον αφορά τις, ε, την τροποποίηση του συντάγματος. διατηρείται πολιτικός ε, τρόπος ε, διορισμού και απομάκρυνσης ε, του Ισαγγελέα Και θα πρέπει σύμφωνα με την Συμφωνία Σύνδεσης με την Ουκρανία να επικυρωθεί η Σύμβαση της Ρώμης. Ε, έχει γίνει η αναβολή όμως της επικύρωσης και παρά αυτές τις προκλήσεις Φαίνεται να έχει γίνει μεγάλο βήμα για την μεταρρύθμιση. Το αν αυτό το βήμα θα είναι βήμα προόδου θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση των αρχών της Ουκρανίας. Θα εξαρτηθεί επίσης από την δική μας ικανότητα να παρακολουθούμε στενά τις διαδικασίες όλες και τη δυνατότητά μας να αγωνιστούμε για το δικαίωμά μας σε δίκαιη δίκη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβασή σας, καθώς επίσης για τη συντομία της. Εξοικονομήσαμε έτσι κάποια λεπτά, τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για να ακούσουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα ήθελα λοιπόν ε, καταρχάς να καλέσω τους ευρωβουλευτές ε, να πάρουν το λόγο στο το επιθυμούν. Βλέπω ότι ο κύριος Σφίχτκα το επιθυμεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χάρηκα πολύ που άκουσα όλες αυτές τις παρουσιάσεις και ενημερώθηκα από αυτά που ακούσαμε. μπορώ πάλι και τώρα να ξαναπιστέψω στη δημοκρατία και στη δύναμη της δημοκρατίας. Είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες που επιθυμούν να ζήσουν σε μια χώρα ελεύθερη και δημοκρατική μπορούν να επιτύχουν το στόχο τους. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία μας αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο Έλμαρ Μπρόκ στην αρχή της συνεδρίασης είπε ότι μια μεταρρύθμιση τέτοιου εύρους σε ένα τόσο σημαντικό τομέα όπως είναι η δικαιοσύνη είναι κάτι πολύτιμο. Σήμερα που βλέπουμε ότι ένα τμήμα της Ουκρανίας είναι υπό παράνομη κατάληψη, όταν βλέπουμε ότι τα εδάφη της έχουν, τα έχει σφετεριστεί κάποια γειτονική χώρα, όταν βλέπουμε τι συμβαίνει στα σύνορα, χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα. Βέβαια αυτά που γίνονται ενέχουν με κάποιο μεγάλο κίνδυνο και είστε πρόθυμοι να τον αναλάβετε αυτόν τον κίνδυνο. Το εύρος αυτών των δράσεων πραγματικά ε, με εκπλήσει και συμφωνώ με τον τελευταίο ομιλητή ότι χρειάζεται χρόνος. Πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτές τις δράσεις να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους. Εγώ δεν θα ήμουν υπέρ ενός συστήματος εκτεταμένου ελέγχου όπου κάποια θεσμικά όργανα θα επιβλέπουν επί μακρόχρονικό διάστημα το δικαστικό σύστημα στην Ουκρανία. Αλλά Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας, πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ουκρανία και ίσως αυτό να είναι και η τελευταία ευκαιρία για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη αυτή. Οι πολίτες πρέπει να θελήσουν την αλλαγή. Τώρα μετά τα σχόλια αυτά έχω και μια ερώτηση. Μιλήσατε για αυτή την ανώτατη επιτροπή η οποία θα επιφορτιστεί με την ε, προετοιμασία του διορισμού των δικαστών. Όσον αφορά τους υποψηφίους, γιατί ε, και εγώ έκανα σπουδές νομικής στο Πόσναν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήμουν καλός υποψήφιος για να γίνω δικαστικός. Για να γίνω δικαστής θα έπρεπε να περάσω από μια μεγάλη σειρά εγκρίσεων ε, και κρίσεων. Εγώ για προσωπικούς λόγους δεν ακολούθησα μια τέτοια πορεία για να γίνω δικαστής. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής όταν θα γίνει η επαλήθευση των στοιχείων των δικαστών από αυτή την Επιτροπή και θα γίνει ο διορισμός τους. Υπάρχει και κάποιο άλλο επίπεδο ελέγχου. Και άλλη μια ερώτηση σχετικά με τον εισαγγελέα. νόμιζα ότι πρόκειται για, μια πολιτική διαδικασία, ένα τομέα που υπάρχει πολιτική επιρροή. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί η διαφθορά ε, πλήττει όλη τη χώρα. Και υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος στο να έχει πολιτικό χαρακτήρα η εισαγγελία. Εμπνέομαι από τα όσα συμβαίνουν στη δική μου χώρα, γι' αυτό τα λέω. Ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες από την εισαγγελία. Θα έχει πολιτικό, προ, ε, πολιτικό χαρακτήρα. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω εξ να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους και να τους ευχηθώ καλή τύχη με την υλοποίηση όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρει η Ουκρανία. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία, όπου ήμουν και Υπουργό Δικαιοσύνη και έχω την εμπειρία μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό τομέα. Περνώντα από ένα δικτατορικό καθεστώ σε ένα δημοκρατικό καθεστώ, είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση αυτή. Και χρειάζεται και μεγάλο χρονικό διάστημα. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να γίνει και γρήγορα γιατί αν προγραμματίσετε να το κάνετε σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, κάποια στιγμή θα χάσετε την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη. Θα θεωρήσουν οι πολίτες ότι δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν θέλω να πω ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι δικαίωμα των πολιτών. Έχουν δικαίωμα σε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη σημαίνει ανεξάρτητη από κυβερνητικές επιρροές, ανεξάρτητη από διαφθορά, γιατί οι δικαστές πρέπει να υπακούν μόνο τον νόμο. Και το λέω γιατί πολλοί δικαστές σε πολλές χώρες που βρίσκονται σε μετάβαση κατάλαβαν ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη σημαίνει ότι είχαν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι ήθελαν και κανεί δεν θα μπορούσε να τους πει κουβέντα. Ανεξαρτησία λοιπόν της δικαιοσύνης σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να χαίρουν ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό όταν ξεκινάτε με τη μεταρρύθμιση ενός δικαστικού συστήματος. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και εμείς είχαμε πολλά προβλήματα στην ε, χώρα μου μέχρι ότου καταλάβαμε ότι έπρεπε να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και έχω μια σχετική ερώτηση. Αν προγραμματίσετε μια ενοποίηση της δικαστικής δικαιοδοσίας και ενοποίηση της νομολογίας, θα είναι χρήσιμο νομίζω γιατί ε, αν ε, οι αποφάσεις διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και ε, για παρόμοια δικήματα οι ποινές είναι από ένα έως τρία χρόνια παραδείγματο χάρη, αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα επειδή σε πολλές χώρες, Κροατία, Βουλγαρία, Ρουμανία, σε όλες τις χώρες της ε, περιφερειάς μας, περάσαμε από τέτοιο στάδιο. Και οι δικαστές πολύ συχνά λένε ότι εγώ είμαι ανεξάρτητος, δεν με νοιάζει τι έκανε ο συνάδελφος δικαστής, εγώ θα δώσω αυτή την απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχετε ένα σχέδιο για την ενοποίηση ε, του δικαστικού σώματος, να μην περάσει την νοοτροπία ότι είμαι ανεξάρτητος και κάνω ό,τι θέλω δεν είναι τυχαία η απονομή δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να εξαρτάται ο πολίτης από το ποιος είναι ο δικαστής. Θα πρέπει να είναι προβλέψιμη η απονομή της δικαιοσύνης. Γι' αυτό χρειάζεται κάποια ενοποίηση. Βεβαίω και μπορεί να διαφοροποιηθεί κάποιος εφόσον υπάρχει κατάλληλη αιτιολόγηση. Ενοποίηση λοιπόν της ε, δικαστικής πρακτικής και δεν υπάρχει πια ε, η διάκριση με, το, με τη Βρετανική νομολογία. Έχουμε κοινό, κοινή νομολογία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χρησιμοποιεί το ε, νομικό προηγούμενο. Το ίδιο κάνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Δεν έχουμε μόνο ε, τον νόμο τον οποίο ερμηνεύουμε, αλλά λαμβάνουμε υπόψη μας και την ομολογία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν έχετε ένα σχέδιο ενοποίησης της ε, νομολογίας και αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με το ότι πρέπει να εξηγήσετε, όπως είπα στην αρχή στους δικαστές, ότι ανεξαρτησία σημαίνει δικαίωμα των πολιτών να έχουν ανεξάρτητη δικαιοσύνη και όχι δικαίωμα των δικαστών να είναι ανεξάρτητοι από τους άλλους και να κάνουν ό,τι θέλουν. Άλλο ένα σχόλιο τώρα. Ο τελευταίος ομιλητής από τη μη κυβερνητική οργάνωση μας είπε ότι οι πολίτες δεν πιστεύουν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις γιατί πιστεύουν ότι θα υπάρξει αμοιβαία συγκάλυψη των δικαστών του δικαστικού σώματος. Είπατε επίσης ότι υπάρχει και αντίσταση των δικαστών. Επιβεβαιώνω ότι όντως θα συμβεί αυτό που λέτε, γιατί αυτό συνέβη και σε όλες τις χώρες που πέρασαν από αντίστοιχη κατάσταση. Η δημιουργία αυτών των δικαστικών συμβουλίων, επιτροπών, ανωτάτων συμβουλίων και ανωτάτων επιτροπών, όπως και να τα λέτε, δίνει εξουσία σε κάποιους δικαστές που αποφασίζουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, αποφασίζουν για τις πειθαρχικές ποινές και θα συγκαλύψουν άλλους δικαστές σε όλες τις χώρες, ε, σχεδόν όλες τα, τουλάχιστον συνέβη αυτό. Και όντως υπάρχει αντίσταση στην αλλαγή πάντοτε, γιατί δεν αρέσει στους ανθρώπους να αλλάζουν τις συνήθειές τους και τα δικτυά τους δεν τους αρέσει να αλλάζουν νόμους γιατί θα πρέπει να τον μάθουν και να αλλάξουν τον τρόπο που εφαρμόζουν τον καινούριο νόμο. Άρα αντίσταση στην αλλαγή υπάρχει και συγκάλυψη θα υπάρχει όπως είπατε. Πρέπει να προσπαθήσετε να το αλλάξετε αυτό και υπάρχουν λύσεις. Μπορείτε να φέρετε και κάποιους που είναι εκτός του, από έξω από το δικαστικό σώμα. Διαφορετικά οι πειθαρχικέ ποινέ δεν θα λειτουργήσουν και δεν θα γίνει εξυγίανση του δικαστικού σώματος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Παρακαλώ. Χαίρομαι που μπορώ να πάρω το λόγο, διότι δεν είμαι μέλος ε, των δύο αυτών επιτροπών. Ε, συμμετέχω όμως ε, στην αντιπροσωπεία προς την Ουκρανία. Γι' αυτό χαίρομαι που μπορώ να πάρω το λόγο. Όλοι γνωρίζουν ότι θέλω μια επιτυχή διαδικασία μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματο στην Ουκρανία. Νομίζω όμω πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά αυτά που είπε η τελευταία ομιλήτρια. ακόμα και αν φαίνεται, αυτά που είπε ο τελευταίος ομιλητής του πάνελ, ε, ακόμα και αν φαίνεται επιτυχής η μεταρρύθμιση για μας εδώ, το κοινό γενικά δεν έχει πιστεί ότι έχουν επιτευχθεί ή ότι θα επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι σύντομοι. Μιλάμε δηλαδή για την ανεξαρτησία των δικαστών από την ε, πολιτική επιρροή και μπορώ να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο κύριος Μπρόκ στο τέλος της παρέμβασής του. Ο φίλος μας, ο κύριος ε, Λουτσέγκο, ήταν ένας από τους ε, πολύ εντυπωσιακού πολιτικούς στο Μαϊντάν και αγωνίστηκε για την ε, δημοκρατία, αλλά η απόφαση να διοριστεί τελικά είχε αρνητική αποδοχή στο πώς βλέπει το κοινό της Ουκρανίας την ιδέα περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Και θα ήθελα να καλέσω τους Ουκρανούς που είναι αρμόδιοι για τις μεταρρυθμίσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτή τη νέα προσπάθεια μεταρρυθμίσεων, να μην κάνουν τα ίδια λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Να θεωρήσουν τους εαυτούς τους καλύτερους πολιτικούς, ε, να είναι κοντά στους θεσμούς του κράτους ε, και έτσι να θεωρούν ότι μπορούν να διασφαλίσουν ε, ότι όλα είναι καλά. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ανεξάρτητους θεσμούς, ανεξάρτητους δηλαδή από την πολιτική επιρροή. Ναι, κοιτώ το ρολόι. Συμφωνώ πάντως με τον τελευταίο μιλητή. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ε, δεν είναι όμως ακόμα απόλυτα πιστική. Ναι, πράγματι έχουμε προβλήματα χρόνου. Ε, η τελευταία παρέμβαση, αν είναι δυνατόν να παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ούτε κι εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή αυτή, είμαι όμως μέλος της αντιπροσωπείας προς την Ουκρανία και με απασχολεί το θέμα αυτό. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Στο πάνελ δεν βλέπουμε τον απλό Ουκρανό τον ταξιτζή, τον μικρό μαγαζάτορα. Έχω πάει πολλές φορές στην Ουκρανία, πριν λίγες εβδομάδες ήμουνα εκεί και βλέπω, ακούω ποια είναι η κοινή γνώμη που θεωρεί ότι η επανάσταση της αξιοπρέπειας ε, κλειδώνησε τις δομές του παρελθόντος, ε, δεν κατάφερε δεν κατάφερε όμως να τις διαλύσει. Διότι η ίδια πολιτική και οικονομική ελίτ κινεί τα νήματα. Και αυτό βέβαια είναι πρόβλημα. Ξέρω ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης εξορισμού είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και ο, χρόνος δεν μας βοηθάει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα είναι εντυπωσιακά. Αλλά όλα αυτά θα, αποτελέσουν, θα απαιτήσουν πολύ χρόνο. Δύο ερωτήσεις έχω. Ο κύριος Μπέλετ είπε ότι ακολουθήθηκαν οι περισσότερες συστάσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπήρχαν συστάσεις που δεν ακολουθήθηκαν, που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν προβλήματα. Υπήρξαν σημαντικές συστάσεις που δεν ακολουθήθηκαν, όπου θα πρέπει να δοθεί η συνέχεια. Και μία ακόμα ερώτηση προς τον κύριο Πετρέγκο ή τον κύριο Φιλάτοφ. Ε, θα υπάρξει αναδιοργάνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου με νέους διαγωνισμούς. Οι υποψήφοι μπορεί να είναι δικαστές, νομικοί, ακόμα και για δικηγόροι. Ποιος φορέας ε, θα εκπονήσει τον, ε, τις ερωτήσεις του διαγωνισμού, θα έχετε διεθνή επιτροπή για να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Σας ευχαριστώ, εξαντλήσαμε το χρόνο μας για τις ερωτήσεις. Δεν έχουμε χρόνο για τις απαντήσεις. Αυτό βέβαια εντάξει δεν μπορεί να γίνει. Ας ξεκινήσω από την κυρία Σιρότη να τη ζητήσω να είναι σύντομη. Θα απαντήσω σύντομα σε όσε ερωτήσει μπορώ και θα δώσω μετά το λόγο στου συναντέρφους. Καταρχά, ε, χαίρομαι που η παρουσίαση του Ρωμάν ήταν αυτή που αναφέρθηκε περισσότερο, διότι έτσι έχουν τα πράγματα. Και χαίρομαι που αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Αυτό είναι πολύ καλό. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και το ανέφεραμε και εμείς. Ε, δεν, δεν υπάρχει πολύ εμπιστοσύνη, υπάρχει όμως ελπίδα. Όσον αφορά την εισαγγελία, ναι, δυστυχώς. Ο διορισμός του εισαγγελέα αποτελεί μέρος του πολιτικού πακέτου. Και πιστεύω ότι αυτό είναι συνέπεια της πολιτικής ανοριμότητας, διότι δεν καταλαβαίνουμε ότι ειδικά η θέση του Γενικού Εισαγγελέα είναι νομική και δεν αποτελεί μέρος του πολιτικού τοπίου. Με όλο το σεβασμό μου προς τον παρόντα Γενικό Εισαγγελέα, τον γνωρίζω από τον Κοινοβούλιο και τον σέβομαι πολύ. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Πρέπει να ξεπεράσουμε όμως τα προβλήματα αυτά. και να φτάσουμε να έχουμε πιο επαγγελματική προσέγγιση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Η μακροπρόθεσμη απόφαση θα ε, είναι η αλλαγή στην νομική εκπαίδευση, διότι μόνο αν ο κόσμος καταλάβει τι είναι το κράτος δικαίου θα μπορέσει να το ακολουθήσει. Και δυστυχώς αυτό απαιτεί μια γενιά. Δεν ξέρω τι γίνεται στις δικές σας χώρες, αλλά στην Ουκρανία ακόμα δεν διδάσκουμε το κράτος δικαίου. Διδάσκουμε τα πρότυπα, τα οποία όμως δεν βοηθούν. Αν κοιτάξουμε το θέμα πιο βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει καταρχάς να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου και ιδιαίτερα όσον αφορά τις απόψεις τους και τα ηθικά πρότυπα. Αυτό το έχουμε συζητήσει. Αφήνω το λόγο στους συναδέρφους να συνεχίσουν. Σας ευχαριστώ κύριε Πετρέγκο. Πολύ σύντομα θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας σχετικά με την ανεξαρτησία των δικαστών μας και του δικαστικού σώματος και τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η ανεξαρτησία των δικαστών είναι δικαίωμα του λαού, δεν είναι δικαίωμα του δικαστή, είναι δικαίωμα της κοινωνίας. Και η απαιτεί υποχρέωση για τον δικαστή να είναι ανεξάρτητος από πολιτικούς, υπουργούς, ε, ε, από χρήμα κλπ. Αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, λόγω του παλιού συντάγματος, όλοι οι δικαστές ήταν υπερβολικά ανεξάρτητοι, είχαν εκτεταμένες ασυλίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσφύγει κανείς στο δικαστήριο ενάντια κάποιου δικαστή, ακόμα και αν έχει σκοτώσει κάποιον στον δρόμο. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία. Και είχαμε κι άλλο ένα πρόβλημα. Ήταν ανεξάρτητη στο πλαίσιο της νομοθεσίας, εξαρτώνταν όμως από ολιγάρχες, κυβερνήσεις, πολιτικούς, χρήματα. Υπήρχε διαφθορά. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Έχουμε όμως τώρα μια πραγματική ευκαιρία και θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας σχετικά με τους διαγωνισμούς και την αναδιοργάνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Δεν αναδιοργανώνουμε το δικαστήριο, δημιουργήσαμε νέο με την ε, τροποποίηση του συντάγματος και με τον εφαρμοστικό νόμο. Δημιουργήσαμε νέο ανώτατο δικαστήριο, νέα εφετεία και μέσα σε τρία χρόνια πρέπει να γίνει αυτό με τα Και οργανώνουμε δημόσιους διαγωνισμούς για όλες τις θέσεις δικαστών σε αυτά τα νέα δικαστήρια. Για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της Ουκρανίας, στους διαγωνισμούς αυτούς μπορούν να συμμετάσχουν όχι μόνο οι δικαστές, Ποιο ήταν το πρόβλημα του συστήματος της Ουκρανίας. Εάν κάποιος ήθελε να είναι δικαστής στο εφετείο έπρεπε να εργάζεται στο τοπικό δικαστήριο. Εάν ήθελε να ε, εργαστεί στο ανώτατο δικαστήριο έπρεπε να περάσει από το εφετείο πρώτα. Ήταν λοιπόν ε, ε, ερμητικά κλειστό το σύστημα. Τώρα λοιπόν το έχουμε ανοίξει. Θέλουμε να δούμε νομικούς νέους από τον ιδιωτικό τομέα, από τα πανεπιστήμια. Και γι' αυτό ε, για τη διαφάνεια των διαγωνισμών αυτών, για, τους διαγωνισμούς αυτούς. Σήμερα είχαμε συνάντηση με την Επίτροπο και σας ζητήσαμε επιρογνώμονες να μας βοηθήσετε να οργανώσουμε αυτούς τους διαγωνισμούς. Εγώ προσωπικά δεν θέλω εξαρτημένους δικαστές. Ήμουνα δικηγόρος όταν έγινε η Επανάσταση και πάλευα ενάντια σε αυτό το σύστημα. Λίγη αξιοπρέπεια ήθελα από τους δικαστές και λίγη ανεξαρτησία από πλευρά τους ε, απέναντι ε, στις υποθέσεις όπου δικάζονταν ε, οι επαναστάτες. Αλλά δεν έγινε αυτό. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να ανανεώσουμε όλο το σύστημα. και έτσι θα έχουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Εφόσον είναι ανεξάρτητο το σύστημα, αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σας ευχαριστώ. Υπήρξε κάποια ερώτηση προς τον κύριο Φίλατοφ. Παρακαλώ, πολύ σύντομα. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Και εγώ θα αναφερθώ στο θέμα της ανεξαρτησίας. Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ σκόπιμη ερώτηση. συζητήσαμε την ισορροπία ανάμεσα στην ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης και, την, ε, και το Σύνταγμα. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει εχέγγυα στο σύστημα και στο Σύνταγμα. Ανεξαρτησία δεν σημαίνει ατιμορρησία δεν σημαίνει πλήρη απουσία ελέγχου και ευθύνη. Με βάση τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, δίνουμε προτεραιότητα στους δικαστές, αλλά στο σώμα αυτό συμμετέχουν και δικηγόροι, νομικοί καθηγητές. Δεδομένων των μηχανισμών ε, για την ε, λήψη αποφάσεων στο σώμα αυτό, πιστεύουμε ότι θα διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ανεξαρτησία και την υπευθυνότητα. Επίσης, ε, όσον αφορά την δικαιοδοσία, την ενοποίηση. Αυτό ήταν ένας από τους στόχου μας κατά τη δημιουργία του νέου ανώτατου δικαστηρίου. Ένας από τους στόχους μας ήταν όλα τα ανώτατα δικαστήρια να ε, ενοποιηθούν για να λύσουμε ακριβώς το πρόβλημα που αναφέρατε. Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με τις συστάσεις που δεν ακολουθήθηκαν, Υπήρχαν κάποια δευτερεύοντα ζητήματα όσον αφορά το Υψηλό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και τον διορισμό του ε, Γενικού Εισαγγελέα. Η σχετική επιτροπή πρότεινε το Κοινοβούλιο να ψηφίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων για να ληφθεί η απόφαση αυτή. Αλλά αυτό στην πράξη θα σήμαινε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προβλήματα όσον αφορά το σχηματισμό του υψηλού Συμβουλίου Δικαιοσύνη και τον διορισμό του Γενικού Εισαγγελέα, διότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί πολιτική συνένεση σε τόσο υψηλό επίπεδο. Μετά λοιπόν από συζητήσεις με την Επιτροπή Μένες, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε άλλη διαδικασία. Αυτές είναι οι δύο μόνες συστάσεις που δεν ακολουθήθηκαν που υπήρχαν στο αρχικό κείμενο. Η άλλη είχε να κάνει με το δικαίωμα του Κοινοβουλίου για ψήφο μη εμπιστοσύνης απέναντι στο Γενικό Εισαγγελέα. Κάτι που οδηγεί στην απόλυσή του. Στο αρχικό κείμενο που συμφωνήθηκε από την Σταγματική Επιτροπή, το Κοινοβούλιο δεν είχε το δικαίωμα αυτό, διότι θεωρήθηκε ότι μπορεί να είναι πολιτικό εργαλείο για να ε, επηρεάζει τη δουλειά του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν θέλαμε όμως το Κοινοβούλιο να έχει κάτι τέτοιο, διότι κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι τελείως μη πολιτικό πρόσωπο ο Γενικός Εισαγγελέας και δεν θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, αλλά με στόχο ε, την εξέβρεση συνένεσης μεταξύ των μελών του Κοινοβουλίου και για να στηρίξουν αυτό το Σύνταγμα, ο Πρόεδρος αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιδέα αυτή. διότι υπήρχε κίνδυνο οι τροπολογίε να μην ε, συμφωνηθούν από το Κοινοβούλιο εφόσον ε, ε, παραμείνει αυτή η προϋπόθεση. Αυτές ήταν οι δύο συστάσεις που δεν ακολουθήθηκαν. Όλες οι άλλες συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο κειμένου. Ευχαριστώ, κύριε Φιλατόφ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Φιλατόφ απάντησε στις ερωτήσει σε σχέση με τι συστάσει. Θέλω μόνο να προσθέσω ότι βρίσκεται λεπτομερεί πληροφορίε στο δικτυακό τόπο τη Επιτροπή τη Βενετία. Κύριε Κοζιακόφ, αν θέλετε να απαντήσετε συντομία και εσεί, θέλω όλου να σα πω να σας καλέσω να, επισκεφθείτε την Επιτροπή της Επιλογής των Δικαστών στη διάρκεια του διαγωνισμού για τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ήδη ε, Στη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαστών χρησιμοποιούμε ε, την ε, νομοθεσία και εδώ σε αυτό το ε, φιλμ που σας ανέφερα μπορείτε να δείτε τι γίνεται ακριβώς. Όταν εγώ μιλώ μπορούν όλοι να με δουν και να με ακούσουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Επιτροπή. Ότι δηλαδή κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έρθει να καθίσει σε μια άλλη αίθουσα όπου αναμεταδίδεται σε απευθείας μετάδοση ό,τι γίνεται στην αίθουσα όπου γίνεται η αξιολόγηση των δικαστών. Θα το συνεχίσουμε λοιπόν αυτό και είστε πρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε τη διαδικασία. Ο κύριος Κουμπίκα. με συγχωρείτε. Τώρα, ε, δύο λόγια για την έλλειψη εμπιστοσύνη. Δεν αφορά μόνο του δικαστέ, αλλά και του πολιτικού και την πολιτική εξουσία. Διότι δύο χρόνια μετά από την επανάσταση τη αξιοπρέπεια. Διότι ε, χωρίς αλλαγή στο Σύνταγμα δεν φάνηκε να λειτουργεί τίποτα καλύτερα. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν εμπιστεύεται το μέλλον. Εμείς τώρα που δουλεύουμε με τις ΜΚΟ μας στον τομέα αυτό, προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο το ωφέλη της δικαστικής μεταρρύθμισης και της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Χάουταλα. Ένα σύντομο σχόλιο από την κυρία Μαγκίνες που είναι αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την υπομονή σας και ευχαριστώ και όλο το πάνελ. Μόλις έφτασα, ήταν εδώ οι συνεργάτες μου. Έχω να κάνω μόνο ένα σχόλιο όσον αφορά τη διεθνή απαγωγή, τις διεθνείς απαγωγές παιδιών. Ε, θέλει εκεί μεγάλη προσοχή και γι' αυτό και ήρθα εδώ για να σας μιλήσω και να ε, ε εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συνεργασία μαζί γιατί έχουμε υποθέσεις ε, που αφορούν αφορά, ε, ε, αφορούν ε, τα παιδιά και τους γονείς παιδιών από μεχτούς γάμους που βρίσκονται είτε στην Ουκρανία είτε στην Ευρώπη είναι πολύ δύσκολο και φυσικά η σωστή και αδιάφθορη διαδικασία είναι πολύ σημαντική για προς του παιδιού, προς το συμφέρον του παιδιού κάθε φορά. Καλή επιτυχία λοιπόν με όλες τις μεταρρυθμίσεις σας. Η κυρία Χάουταλα τώρα που είναι συν πρόεδρος της ε, συνέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας να ε, μας πει ε, τα συμπεράσματά της. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κανεί δεν ήρθε εδώ για να τον επενέσουμε και να του πούμε ότι όλα πάνε τέλεια. Ε, το ξέρω, δεν είστε εδώ γι' αυτό, ούτε και εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό, αλλά είμαι ωστόσο ευτυχής που μπορέσατε να, να κάνετε αυτή την προσπάθεια. Όλοι υποστηρίζουμε τη δουλειά αυτή, ώστε όντως να εξυγχρονιστεί το δικαστικό σύστημα και να ανεξαρτητοποιηθεί και είναι μεγάλη μου χαρά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις διάφορα, τα διάφορα σώματα, την αντιπροσωπεία με την Ουκρανία και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων συνεργάζονται πραγματικά για να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες. Απλά θυμάμαι μια ε, ιστορία από τη Φιλανδία, αυτό το ρητό που λέει ότι φαίνεται, ε, αυτό που είναι φαίνεται. Ε, και κάποτε αποκαλύφθηκε ότι η διεύθυνση email του Γενικού Εισαγγελία της Φιλανδίας είχε ακριβώς την ίδια διεύθυνση όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και, το, και άλλαξε αυτό για να φανεί ότι δεν υπάρχει λόγος να σκεφτεί κανείς ότι υπήρχε συσχέτιση και, ή μάλλον σχέση, εξάρτηση ε, με, από, του Γενικού Εισαγγελέα από το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Πολύ μικρές λεπτομέρειες μπορεί να δώσουν λαβή για υποψίες και καχυποψία γενικά. Για να βάλουμε λοιπόν σε μια κάποια προοπτική όλη αυτή τη συζήτηση, θέλω να κάνω δύο γενικές παρατηρήσεις. καταρχά, επειδή ε, προέρχεστε από την ε, σοβιετική κληρονομιά, έχετε προχωρήσει πιστεύω πάρα πολύ και επειδή η Ουκρανία είναι τόσο τεράστια χώρα, μόνο και μόνο ο αριθμός των δικαστών, 8.000 δικαστές μας είπατε, είναι εντυπωσιακό αριθμός. Αλλά όπως είπε και η κυρία Μακοβέη που είναι από τη Ρουμανία, δεν είναι εύκολη η μεταρρύθμιση ενός δικαστικού σώματος που με τόσο βαριά μάλιστα κληρονομιά. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε στο όλα να γίνουν πολύ συστηματικά και ο κύριος Στομπίνσκι ήταν εδώ και μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά προσπαθεί να βοηθήσει με εμπειρογνωμοσύνη. Όπως είπε και ο Υπουργός, ε, Οι παρατηρήσεις ε, των πολιτών, ωστόσο, θα πρέπει πάντοτε να μας κάνουν να σκεφτούμε ε, και ένα από τα σοβαρότερα στοιχεία για μεταρρυθμίσει σε χώρε όπω η Ουκρανία, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Μολδόβα, που επίσης ε, τις προσέχουμε πάρα πολύ. Σημαντικό είναι η κοινωνία των πολιτών να μπορεί να σχολιάσει και να επικρίνει και να συμβουλέψει κάποιε φορέ την κυβέρνηση ακόμα και το Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν πραγματικά ότι οι επικρίσεις αυτές θα θεωρηθούν ως επικοδομητική συμβολή προς όλη αυτή την προσπάθεια. Κάτι το οποίο παρατηρώ είναι πως δυστυχώς η κύρωση του καταστατικού της Ρώμης για να μπείτε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει καθυστερήσει γιατί αυτό δεν είναι προς το συμφέρον μιας χώρας που έχει που είναι στόχος ε, στρατιωτικής ε, επίθεσης από πλευρά της Ρωσίας που επίσης έχει συχνά κατηγορηθεί για παραβιάσεις ε, το διεθνούς ποινικού δικαίου. Θα ήταν καλό λοιπόν να γίνει πιο γρήγορα. Κανεί δεν το ανέφερε, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω λοιπόν πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επικεντρώνει τις προσπάθειες του στη συνεργασία με την Κομισιόν για να σας στηρίξουμε σε, αυτό, αυτή την προσπάθεια. Εδώ λοιπόν ήταν μια δοκιμή για να δούμε πώς μια τέτοια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μπορούν, μπορεί να βοηθήσει. Θα υπάρξουν και άλλες δυνατότητες για άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου να στηρίξουν τις προσπάθειες της οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που και ελπίζω και ότι από την πλευρά της ε, Συνέλευση Euronest θα το στηρίξουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητέ σε αυτό το πρώτο γύρο που ήρθατε και πάλι θα αλλάξουμε θέσεις. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Λουτσέγκο, τον κύριο Λάτσιγκας και τον κύριο Σάμπονιν να έρθουν εδώ για το δεύτερο πάνελ.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 Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο γύρο της συζήτησης, μεταρρύθμιση της ε, υπηρεσίας του Γενικού Εισαγγελέα και θα δώσω το λόγο στο φίλο Γιούρι Λουτσένκο που είναι Γενικός εισαγγελέα της Ουκρανίας. Δέκα λεπτά για τον κύριο Λουτσένκο. Θα έρθει και ο Υπουργός, αλλά έχει ήδη λάβει το λόγο, οπότε θα κάνουμε λίγο εξοικονόμηση χρόνου. Κύριε Λουτσένκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πονκρίτς. Θα μιλήσω ουκρανικά. Сьогодні вже про це говорилося, але я завжди починаю свої. Θέλω ε, να πω, όπως λέω πάντοτε ξεκινώντας τις ε, ομιλίες μου σε ξένες χώρες, ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου. Η Ουκρανία είναι σε πόλεμη κατάσταση όχι μόνο λόγω του πολέμου με τη Ρωσία, αλλά και γιατί καταπολεμά την συστημική διαφθορά και εγκληματικότητα που ε, είναι γνώρισμα της χώρας από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. προηγούμενοι ηγέτες της χώρας δημιούργησαν μια κρατική μαφία όπου όλα, όλοι οι θεσμοί δούλευαν για τη μαφία της οικογένειας του Γιαννουκόβιτς. Εγώ έφτασα στο κοινοβούλιο μετά το δεύτερο Μαϊντάν ως ε, επικεφαλής της μεγαλύτερης ομάδας στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο και σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε αλλάξει πολλά στην νομοθεσία μας και τώρα, κατά τη γνώμη μου, η Ουκρανία έχει την πιο αυστηρή νομοθεσία κατά της διαφθοράς στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Την περασμένη εβδομάδα ξεκινήσαμε την ε, πιο ριζική μεταρρύθμιση με την υποστήριξη της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου. Στη Γενική Εισαγγελία είχαμε τρεις νέους γενικούς εισαγγελείς, αλλά παραμένει ε, φέουδο της ε, Σοβιετικής κυριαρχίας. Δεν θα μπορούσε κανείς να συνηθίσει ε, αυτά τα οποία βλέπουμε στην εισαγγελία για τον τρόπο ζωής και το ύφος άσκηση των καθηκόντων των εισαγγελέων. Πρέπει να τονίσω ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε καμία ευθύνη για τους εισαγγελείς. Κανένας εισαγγελέας δεν έφερε ευθύνη για τις πράξεις του. Αυτό το αλλάξαμε. Ε, τι να σας πω, ότι ε, κάποιος σε οδικό ατύχη, σε τροχαίο ατύχημα σκότωσε έναν άνθρωπο και συνέχισε να είναι εισαγγελέα. Εγώ αντικατέστησα τρεις εισαγγελείς ένας είναι ε, πρώην διπλωμάτης ε, και άλλος ένας ε, νομικός. Και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία. Για το 2016 είναι ξεκάθαρα τα καθήκοντα που έχουμε θέσει για το έργο μας. Θέλουμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, να κάνουμε πλήρη εκαθάριση του συστήματος. Το πρώτο βήμα θα είναι το εξής, να συγκρίνουμε την διακήρυξη ακαιρεότητας του εισαγγελέα με το εισόδημα της οικογένειάς του. Ε, αναθέσαμε σε έναν 30 30χρονο συνάδελφο αυτό το έργο, κάποιον που ήρθε από ε, ε, τη Γαλλία που ήρθε και πολέμησε για την Ουκρανία, έχισε το αίμα του για την Ουκρανία και θα συνεχίσει να αγωνίζεται κατά της διαφθοράς. Δεύτερο βήμα θα είναι να έχουμε νέα πρόσωπα στην Γενική Εισαγγελία. Τρίτο βήμα θα είναι να δημιουργήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών με το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητού που θα ασχολείται με έρευνα και ανάκριση για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της εισαγγελίας. Το δεύτερο σημαντικό μας έργο είναι ότι πρέπει τα μεγάλα ψάρια να πιαστούν. Πρέπει να δείξουμε ότι στρεφόμαστε κατά των ε, μεγάλων ψαριών. Μίλησα για την μαφία του κυρίου Γιαννουκόβιτς και δεν πρέπει να φοβόμαστε να το λέμε. Η δική του περίπτωση είναι μοναδική, διότι από την πρώτη μέρα ε, της εξουσίας του άσκησε πιέσεις στο συνταγματικό δικαστήριο. Υπέγραψε ε, προδοτικές συμφωνίες με την Ρωσία, επιτρέποντάς τους να φέρουν στρατιωτικές μονάδες στην Κρυμαία που οδήγησαν στην προσάρτησή της. Δημιούργησε ε, ευκαιρίες για να ανθίσει η διαφθορά στη χώρα μας με απάτες που έφταναν τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια η κάθε απάτη. Ό,τι και να κέρδιζε το κράτος, τα μισά πήγαιναν στις τσέπες της οικογένειας Γιανουκόβιτς. Και πολύ λίγα έμεναν για το κρατικό προϋπολογισμό. Όλα αυτά καταράκωσαν τον εθνικό προϋπολογισμό. Ο Γιαννουκόβιτς δανειζόταν από το Κρεμλίνο με αντάλλαγμα την Ουκρανική κυριαρχία. μια σειρά εγκλημάτων και τέλος ζήτησε ο Γιαννουκόβιτς από τον πρόεδρο Πούτιν να φέρει τα στρατεύματά του στην Ουκρανία. Και θα συνεχίζουμε να κατηγορούμε τον Γιάννου Κόβιτς ε, γι' αυτό. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα ασχολούμεθα μόνο με τα όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά το να ε, αποδώσουμε δικαιοσύνη και να ε, κατηγορήσουμε αυτούς οι οποίοι είναι υπέτοιοι παραμένει βασικό μας καθήκον. θα πρέπει στην ε, Γενική Εισαγγελία να έχουμε εκπροσώπους ε, της νέας γενιάς καθαρών εισαγγελέων. Και να σας πω και κάτι ακόμη, ότι ε, έχουμε μια υπόθεση ενός ατόμου που ήταν στη φυλακή 4,5 χρόνια ε, χωρίς να έχει δικαστεί. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει 12-13 χρόνια στη φυλακή πριν δικαστούν. Θα πρέπει το σοφρονιστικό μας σύστημα να είναι ανεξάρτητο και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. για τα επόμενα χρόνια να σας πω καταρχήν ότι στο, στην οθόνη βλέπετε ε, τις αρμοδιότητες όπως κατανέμονται στο σύστημά μας. Είναι ένα σύστημα παρόμοιο με το αμερικανικό. Μας το πρότειναν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες χώρες. Έχουμε λοιπόν το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητού και ήδη από τον Αύγουστο θα αρχίζουμε να επανδρώνουμε το γραφείο αυτού του επιθεωρητού. Για τα επόμενα χρόνια θέλουμε ε, να επιφέρουμε συστημικές αλλαγές στην εισαγγελία. Θέλουμε να ισχύουν διαγωνισμοί για όλες τις θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα Θέλουμε νέα πρόσωπα, μια νέα κουλτούρα, μια κουλτούρα συνεργασίας. και θα μπορούν νέοι άνθρωποι ε, να ανελιχθούν με βάση τα προσόντα τους. Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στο παλιό σοβιετικό σύστημα να επιβάλλει την προσέγγιση του. Θέλουμε νέα πρόσωπα που θα προσληφθούν με βάση νέους διαγωνισμούς και θα μπορέσουν να διοικήσουν σωστά την εισαγγελία. Ε, ε, ξέρω ότι ότι ε, οι εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα για ανάκριση θα ισχύουν μόνο για δύο χρόνια ακόμη και ήμουν και εγώ από αυτούς που το ψήφισαν ε, στο Κοινοβούλιο. Η απόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία. Δεν θα υπάρχει δηλαδή ερευνητική λειτουργία στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Όλα αυτά είναι μεταρρυθμίσεις που όταν ολοκληρωθούν θα έχει ολοκληρωθεί και το δικό μου έργο. θέλουμε να διαχωρίσουμε το έργο του εισαγγελέα από το έργο του ανακριτού και ερευνητού, γιατί είναι επικίνδυνο να συνδυάζονται τα δύο. Η έρευνα και η ανάκριση δεν είναι έργο του εισαγγελέα. Σε μια ομιλία μου στο Κοινοβούλιο, είπα ανοιχτά ότι δεν ήμουν ικανοποιημένος με την αλλαγή ε, του νόμου για την θέση του Γενικού Εισαγγελέα, γιατί επελέγην εγώ που δεν έχω νομική παιδεία. Ήμουν τέσσερα χρόνια στο Υπουργείο Εσωτερικών και δύο χρόνια στη φυλακή ως πολιτικός κρατούμενος. Αυτή ήταν η βάση για την επιλογή μου. Όμως, μην ξεχνάτε ότι με έβαλαν φυλακή υπέρ επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Κάποιος πρέπει να σπάσει αυτό τον κλειό της εξωτερικής διαχείρισης. Και γι' αυτό χρειάζεται κάποιος με πολιτική βαρύτητα για να αλλάξει την ισχύουσα κατάσταση. Αυτό πιστεύουμε ότι θα αλλάξει το σύστημα και γι' αυτό με διόρισαν ώστε να διασφαλίσω νέα πρόσωπα, ανέλυξη με βάση την αξιοκρατία και ε, καταδίκη των προηγουμένων όταν θεωρήσουμε ότι έπραξαν κάτι παράνομο. Την επόμενη φορά που θα είμαι εδώ για να σας μιλήσω θα σας δείξω πια τα αποτελέσματα που θα έχουμε επιτύχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και δίνω τώρα το λόγο στον Κεστού της Λαντσίνσκας, επικεφαλής ε, της Συμβουλευτικής Αποστολής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς την Ουκρανία. Πολλέ προσδοκίε υπάρχουν και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από την πλευρά τη Ουκρανία. Παρακαλώ να προσπαθήσετε να παραμείνετε εντό του δεκαλέπτου. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κυρίε και κύριοι, έχουν γίνει σημαντικέ εξελίξει τα, τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία πριν μόλις ε, μία εβδομάδα οι τελευταίες συνταγματικές ε, τροποποιήσεις σχετικά με το δικαστικό σύστημα υιοθετηθήκαν ε, και τον περασμένο Ιούλιο είχαμε το νέο νόμο για τον Γενικό Εισαγγελέα. Έχουν γίνει τα πρώτα βήματα όσον αφορά την μεταρρύθμιση και υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Ωστέσο, για να υπάρξει πραγματική μεταρρύθμιση, πρέπει να θεωρηθεί ανεξάρτητο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό το εισαγγελικό σύστημα από το κοινό. Κάποια βήματα έχουν γίνει για να γίνει πιο ανεξάρτητο το σύστημα αυτό. Για παράδειγμα, ε, μια διαδικασία ε, επανεπιλογής για όλους τους ε, εισαγγελείς που ξεκίνησε πέρσι. Και η η Συμβουλευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με μη κυβερνητικές οργανώσεις έχει παρακολουθήσει τις διαδικασίες αυτές και διαπιστώνει ότι έχει σημειωθεί η πρόοδος, μόνο δεν έχει ληφθεί η, τελευταία, η τελική απόφαση για την πρόσληψη των ε, εισαγγελέων. Ε, όσον αφορά την ανεξαρτησία, ε, έχουν αναλυφθεί βήματα για να γίνουν έλεγχοι ακαιρεότητα των εισαγγελέων. Ε, θα δοθεί συνέχεια στη διαδικασία αυτή, διότι όπω γνωρίζετε, είναι και αυτό ένα θέμα που βρίσκεται στο θεματολόγιο μεταρρύθμιση του νέου Γενικού Εισαγγελέα. Η αποστολή λοιπόν συνεχίζει να εξετάζει το θέμα. Άλλο θέμα είναι η λογοδοσία απέναντι στο κοινό οι εισαγγελεί ε, θα πρέπει να μπορούν να εξηγούν τις αποφάσεις που λαμβάνουν με βάση το κράτος δικαίου. Και μόνο με βάση αυτό ο εισαγγελέα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Ε, η λογοδοσία βλέπουμε ότι βελτιώνεται. Έχει ξεκινήσει και ποινική δίωξη για 7 ε, περιπτώσεις διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Όπως ανέφερα, ε, έχει τροποποιηθεί το νομικό πλαίσιο, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν. Θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την διερεύνηση μικρών παραπτωμάτων. Δηλαδή ε, οι μικροκλοπές από ε, καταστήματα δεν θα πρέπει να ακολουθούν την ίδια διαδικασία με ε, τις δολοφονίες. Η απλοποίηση της διαδικασίας σημαίνει ότι οι εισαγγελείς μπορούν να επικεντρωθούν στα πιο σοβαρά εγκλήματα. όπως είναι η απάτη και άλλα εγκλήματα. Ε, θεωρούμε ότι πολλά πρέπει να γίνουν ώστε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα να είναι το μέρος όπου θα ξεκινούν οι διαδικασίες αυτές όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στην εισαγγελία και τις αρχές επιβολής του νόμου. Εμείς ε, η αποστολή συμπροεδρεύουμε σε μια ομάδα εργασίας με την Εθνική Αστυνομία και έχουμε καλέσει το Γραφείο του Εισαγγελέα να συμμετάσχει στις εργασίες αυτής της ομάδας εργασίας και χαιρόμαστε που έχουμε ήδη προφορική συμφωνία πάνω στο θέμα αυτό. Στις ε, ποινικέ έρευνες ε, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουμε την Εθνική Αστυνομία, έχουμε το Εθνικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς ε, και σύντομα θα έχουμε και ειδικό γραφείο ερευνών. Σημαντική πρόκληση είναι να διασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αυτών φορέων. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, πολλά βήματα έχουν γίνει ή έχουν προγραμματιστεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο νέος Γενικός Εισαγγελέας θέλει να αναπτύξει ένα σύστημα διαχείρισης των υποθέσεων, ηλεκτρονικό σύστημα και εμείς η αποστολή τον στηρίζουμε στο θέμα αυτό. Κλείνοντας την ομιλία μου θα ήθελα να πω ότι είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε την εισαγγελία της Ουκρανίας σε όλα τα επίπεδα, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να είναι ανεξάρτητη εισαγγελία, ε, ε, αξιόπιστη και αποτελεσματική. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά ως εταίροι. Μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα καθότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές 28 κρατών μελών. Ωστόσο, όσον αφορά την αύξηση της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας, αυτό αποτελεί ένα γενικότερο έργο το οποίο θα πρέπει να αναλάβει η εισαγγελία. Αλλά εναπόκειται και σε μεμονωμένους και στον κάθε εισαγγελέα να αγκαλιάσει αυτές τις αξίες του κράτους δικαίου. Όπως είπε και ένας από τους προαναλύσαντες, ε, οι μεταρρυθμίσεις ε, είναι μακρύς δρόμος. Όλες οι μεταρρυθμίσεις όμως εξαρτώνται τελικά από το λαό. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ κύριε Λευσίνσκας. Δίνω το λόγο στον κύριο Βιτάλη Σαμπούνιν από το σχέδιο δράση κατά τη διαφθορά. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μην μιλήσω ουκρανικά. Καταρχάν, Σας ευχαριστώ όλους καταρχάς για το τι κάνατε για τη χώρα μου. Η ισχυρή σας ε, και σταθερή θέση μας βοήθησε πολύ και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τομπίνσκι του οποίου η φωνή ήταν πραγματική επιρροή στην ε, Ουκρανία και μας βοήθησε επίσης πολύ. Με τη δική σας βοήθεια με την διεθνή στήριξη καταφέραμε τόσα πολλά στην Ουκρανία, αλλά έχουμε ακόμα κάποια πράγματα. Νομίζω πως ε, Μόνο στην Ευρώπη μπορεί κανείς να βρει τόσες πληροφορίες σε σχέση με την ιδιοκτησία ε, ε, και έχουμε το πρώτο μητρό ε, ε, ε, ιδιοκτησιών. Χάρη στη δική σας βοήθεια έγινε αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πετρέγκο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δεν μπορούσε να γίνει χωρίς την προσπάθειά του. Δημιουργήθηκε ένας παράδεισος για τους δημοσιογράφους έρευνας. Όλοι μπορούν να βρουν τα πάντα για όλους. Αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό. Το αποτέλεσμα είναι οι ποινικέ υποθέσει. Ακόμα και εκεί κάναμε μεγάλα βήματα. Έχουμε ένα νέο. Ε, μια νέα επιτροπή που εργάζεται κατά τη διαφθορά στην Ουκρανία και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και λίγα αποτελέσματα έχουμε ήδη, γιατί ο πρώτο ήμιση της θητείας τους μπόρεσαν να πιάσουν δυο φορές περισσότερους δικαστές από ότι το δικαστικό, το, το, το, δικαστικό σύστημα τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Έχουμε το μέλλον, το, έχουμε τον, την, υπο, υπο έρευνα των επικεφαλής της ε, Επιτροπής κατά τη Διαφθοράς, τον πρώην Υπουργό ε, επίσης. Πριν από δύο χρόνια κανείς δεν μπορούσε καν να το σκεφτεί ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Και τώρα έγινε. Το όμως το σύστημα αντιδρά. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι της πολιτικής ελίτ της Ουκρανίας αντιδρά. Προσπαθεί να περικόψει τα κονδύλια για τις νέες αυτές υπηρεσίες. Προσπαθούν να μειώσουν ε, την, ε, το κύρος τους, τις εξουσίες τους δεν θέλουν να αφήσουν ειδικά εργαλεία, ειδικά μέσα, όπως ας πούμε το εισαγγελικό γραφείο να μεταρρυθμιστεί για να μπορέσει να λειτουργήσει. Επίσης, η Επιτροπή κατά Διαφοράς δεν έχει νομικό δικαίωμα να δώσει, να προσφέρει ε, δεν μπορεί να έχει ε, όπλα. Ε, ελαφριά όπλα είναι οι Ουκρανοί δικαστές τόσο επαγγελματίες που μπορούν να, κλείσουν, να σκοτώσουν ακριβώς πριν να γίνει η δίκη σκοτώσουν μάρτυρε. Να σα δώσω κάποια παραδείγματα. Η ευκολότερη έρευνα που μπορούσε να γίνει είναι ένα δικαστή που παίρνει ε, φακελάκια. Βγαίνει, σκάει υπόθεση. Τι κάνει, σκοτώνει το μάρτυρα. Απλούστατο. Τρεις ε, μήνες αφού έστειλε η Ναμπού, η Ειδική ε, Επιτροπή την υπόθεση στο δικαστήριο, η, δίκη δεν ξεκίνησε καν. Οι δικαστέ πετούσαν την υπόθεση από τον ένα στον άλλον. Τρει μήνες, τρία δικαστήρια ολόκληρα άλλαξαν και δεν ξεκίνησε η υπόθεση, η εξέταση τη υπόθεση. Άλλε υποθέσει ε, έρευνα για το μεγαλύτερη κρατική εταιρεία στην Ουκρανία, την Οντέσα, ε, το, εν πάση περιπτώσει μου διαφεύγει το όνομα. Λοιπόν, έγινε μια έρευνα ε, Φανταστείτε τώρα. Το δικαστήριο έβγαλε χωριστή απόφαση ότι αυτό το συγκεκριμένο έντυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο. Αποφάσισε και διέταξε. Ένα σωρό τέτοια παραδείγματα υπάρχουν. Όλο αυτό το σύστημα λοιπόν δεν θα λειτουργήσει εάν δεν αλλάξει η δικαιοσύνη. Και αυτό δεν θα γίνει και δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όσο οι συνάδελφοι. Δεν θα τα καταφέρουμε τουλάχιστον πριν δύο-τρία χρόνια. Λόγω της διαδικασίας. σε πολύ σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς ε, δεν έχουμε καν αυτά τα τρία χρόνια στη διάθεσή μας. Επιπλέον οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην εφαρμοστική νομοθεσία δίνει περισσότερες δυνατότητες ώστε οι, οι παλιοί δικαστές να μείνουν δεν είμαι βέβαιο ότι θα μπορέσουμε, βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να αλλάξουμε όλο το σύστημα, ειδικά στις υποθέσεις κατά της διαφθοράς που είναι τόσο σημαντικές για την πολιτική ελίτ. Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει ένας τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Η δημιουργία νέων δικαστηριών κατά της διαφθοράς. Έχουμε εδώ την, ένα, ένα σύστημα. Θα πρέπει ένα νέο δικαστήριο με χωριστή διαδικασία ε, για επιλογή των δικαστών να φτιαχτεί. Με μια διαδικασία που να μπορούμε, μπορεί να ελέγχεται. Δεν καταλαβαίνω ποια επιρροή, απίστευτη επιρροή μπορεί να υπάρξει για την επιλογή των νέων δικαστών και την εφαρμοστική διαδικασία. Η απόφαση μιας ΜΚΟ ενό ανεξάρτητου σώματο μπορεί να ληφθεί υπόψη, πράγμα που δεν σημαίνει τίποτα στην πραγματική ζωή. Όταν μιλάμε δηλαδή για πολιτικές υποθέσεις, θέλουμε να έχουμε ένα χωριστό δικαστήριο. Ε, χωριστό δικαστήριο για τις υποθέσεις διαφθοράς. And now I should be Επίσης, αυτό το νέο δικαστήριο κατά τη διαφθοράς και την εφαρμοστική νομοθεσία αυτό με την προϋπόθεση να στηθεί ένα τέτοιο δικαστήριο. Χρειάζεται άλλη νομοθεσία ώστε να στηθεί ένα τέτοιο δικαστήριο και μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι ότου να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε τη βοήθειά σας. Βοηθήστε μας όπως ε, μας έχετε βοηθήσει και πριν για να ξεπεράσουμε την πολιτική αντίσταση εντός της Ουκρανίας. Ε, για να μπορέσουμε να στήσουμε ένα τέτοιο δικαστήριο κατά τη διαφθοράς. Γιατί είναι η αντίστροφη μέτρηση για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το νέο σύστημα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Μόνικα Μακοβέη για να κάνει μια παρέμβαση όχι παραπάνω από 10 λεπτά, αναφερόμενη και στις ομιλίες που έγιναν από τα μέλη του πάνελ. Ευχαριστώ. Όπως είπα προηγουμένως και στη Ρουμανία κάναμε μια παρόμοια διαδικασία μεταρρυθμίσεων πριν ενταχθεί η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Um, Και παρατηρώ ότι τα πράγματα είναι παρόμοια. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι σε ένα χρόνο θα ήθελα να τα ξαναπούμε και να δούμε ότι έχετε εφαρμόσει τουλάχιστον τα μισά από αυτά τα οποία μας είπατε, γιατί η υλοποίηση είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, θα συναντήσετε μεγάλη αντίσταση. Η ψήφιση των νόμων είναι το πρώτο βήμα, αλλά είναι και το πιο εύκολο. Θέλετε να κάνετε λοιπόν εξυγίανση του δικαστικού σώματος. Αν το καταφέρετε αυτό, το δικαστικό σώμα θα κάνει την εξυγίανση όλων των άλλων, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών. Επομένως, προτεραιότητα στο δικαστικό σώμα. Αύξηση μισθών για τους δικαστές είναι πολύ σημαντικό και το κάνατε, αλλά δεν αρκεί. Δεν σημαίνει ότι δεν θα παίρνουν δωροδοκίες. Όταν είναι διορισμένοι διαβίου, αυτό είναι καλό γιατί εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους, αλλά ούτε και αυτό αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα είναι διεφθαρμένοι. Αυτό που έχω παρατηρήσει σε πολλές χώρες στην περιφέρειά μας είναι ότι αυξάνονται οι δωροδοκίες και δωροληψίες. Λέτε ότι φαίνεται καινούριου ανθρώπους από τη νέα γενιά. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι τα νέα πρόσωπα από την καινούργια γενιά θέλει περισσότερα χρήματα από την παλαιότερη γενιά. Υπάρχουν περιπτώσεις νέων δικαστών που ζητάνε χιλιάδες ευρώ, μάλλον εκατοντάδες χιλιάδων, ενώ πριν ζητούσαν εκατοντάδες ευρώ, τώρα ζητούν εκατοντάδε χιλιάδων ευρώ. Επομένως δεν είναι η μόνη λύση. Και αν έχετε ε, παραγραφή αδικημάτων ε, μπορεί να μην ε, γίνεται αποδεκτή μια υπόθεση σε ένα δικαστήριο γιατί έχει φτάσει η ημερομηνία της παραγραφής και βλέπετε ότι ο δικαστής δεν έκανε τίποτα. Αν το δείτε αυτό, μπορείτε να εφαρμόσετε πειθαρχική διαδικασία και να τον βγάλετε από το δικαστή, διότι άφησε να παραγραφεί μια υπόθεση. Δεν δημοσιεύει μια υπόθεση, τον διώχνετε. Δεν ε, αιτιολογεί επαρκώ μια υπόθεση, τον διώχνετε. Δηλαδή να προσπαθήσετε να του ε, αποπέμψετε με όλε αυτέ τι μεθόδου, γιατί η εξυγίανση του δικαστικού σώματο είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεύτερο σημείο, η καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό που είπατε μου άρεσε πάρα πολύ. ότι οι πολιτικοί αντεπιτίθενται. Το πιο σημαντικό είναι να γίνει η του πολιτικού σώματος, να καταπολεμήσετε την πολιτική διαφθορά, να κυνηγήσετε τα μεγάλα ψάρια όπως είπατε. Όλες ε, οι υποψήφιες χώρες έχουν αυτό τον όρο, αυτή την προϋπόθεση που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Ένα άλλο σχόλιο που άκουσα είναι ότι θέλετε να καταδιώξετε τα μεγάλα ψάρια, ε, την κρατική μαφία του Κόβιτς. Το να ε, στραφείτε κατά των προηγουμένων δεν αποκαθιστά την εμπιστοσύνη. Δεν λέω ότι δεν έκαναν εγκλήματα, αλλά δεν αρκεί για να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη, γιατί όπου υπάρχει εξουσία και χρήμα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διαφθοράς θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη στο δικαστικό σώμα ή στους πολιτικούς όταν δουν ότι αυτοί που έχουν σήμερα την εξουσία υφίστανται επίσης έρευνα. Ερευνώνται και οι έχοντες τώρα την εξουσία. Στην Ρουμανία δημιουργήσαμε ένα γραφείο εισαγγελέως κατά της διαφθοράς που λειτουργεί πολύ σωστά και εξετάστηκαν και πολλοί υπουργοί και βουλευτές εν ενεργεία και ε, δικαστές ε, και εισαγγελείς. Ήμουν υπουργό ε, στην κυβέρνηση και υπήρχε υπόθεση του αναπληρωτή πρωθυπουργού και βγήκε στα μέσα ενημέρωσης ότι το Γραφείο Εισαγγελέως κατά της διαφθοράς εξετάζει τον ε, ε, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και μου είπε ο Πρωθυπουργό, μα εγώ νόμιζα ότι κατά της αντιπολίτευσης θα στραφείς και του είπα όχι δεν στρέφομαι κατά της αντιπολίτευσης δεν στρέφομαι κατά κανενός εξαρτάται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. οποιοδήποτε συμπεριλαμβανομένης και της ε, κυβέρνησης που έχει τώρα την εξουσία θα πρέπει να ερευνηθεί, θα πρέπει όλοι να ερευνώνται για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Παραδέχομαι ότι η αντιπολίτευση ε, έκανε πολλά αδικήματα. Αλλά αν δεν στραφείτε και κατά των ε, εχόντων την εξουσία όταν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, δεν θα υπάρξει εμπιστοσύνη από τους πολίτες. Τώρα για το σχόλιο σας ότι αντεπιτίθενται οι πολιτικοί. Όταν καταπολεμούμε την πολιτική διαφθορά είναι λίγο παράδοξο διότι θεσπίζουμε νόμους και ζητάμε από τους πολιτικούς να τους ψηφίσουν και ξέρουν ότι αν υλοποιηθούν αυτοί οι νόμοι θα τους δημιουργηθούν προβλήματα, μπορεί και να πάνε φυλακή, μπορεί να τους δημευθεί η περιουσία κλπ. Μπορεί να γίνει λοιπόν σε περίοδο πρώτης ένταξης ή σε περίοδο όπου υπάρχει πίεση, πίεση από την κοινή γνώμη και πίεση απ' έξω. Χρειάζεται δηλαδή να τεθούν κάποια προαπαιτούμενα ως πίεση για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και θα ε, εγκρίνουν η πολιτική την νομοθεσία ελπίζοντας ότι δεν θα υλοποιηθεί και κατά την υλοποίηση θα προσπαθήσουν συνεχώς να, να αντεπιτίθενται. Σε όλες τις χώρες το είδαμε. Στη Σλοβενία, παραδείγματος χάρη, μόλις εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπάθησαν να καταργήσουν ε, την, ε, τον φορέα κατά της διαφθοράς δύο φορές και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση το προσπάθησε και στη Ρουμανία προσπάθησαν να μειώσουν τις εξουσίες ε, αυτού του φορέα κατά της διαφθοράς, προσπάθησαν να αλλάξουν ε, τον νόμο, προσπάθησαν να αποφύγουν την υλοποίηση του νόμου. Δεν θα σταματήσουν οι πολιτικοί. Ε, αυτοί που είναι διαφθαρμένοι δεν θέλουν να σταματήσουν να είναι διαφθαρμένοι, θέλουν να εμποδίσουν τη λειτουργία της αρχής πάταξης της διαφθοράς. Και αν δεν τα καταφέρουν, στη Ρουμανία δεν τα κατάφεραν μετά από 8 χρόνια βάζουν καινούργιες, αρχίζουν καινούργιες μάχες, ότι δεν θα έπρεπε να είναι έγκλημα η σύγκρουση συμφερόντων, γιατί πολλοί έχουν καταδικαστεί για σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί να μην είναι αδίκημα η σύγκρουση συμφερόντων. Συνεχώς λοιπόν προσπαθούν να αντεπιτεθούν και συνεχώς επαγρυπνούμε. Και κάποιοι άνθρωποι σαν εσάς, στις θέσεις που βρίσκεστε εσείς, πρέπει να κρατάτε στεναρή αντίθεση. Όπως είπα και εγώ, όχι στον Πρωθυπουργό. Και δεν είναι εύκολο να λέει κανείς όχι στο αφεντικό του. Βέβαια τα αφεντικά μας δεν είναι συνηθισμένα να τους λέμε όχι, γιατί κανείς δεν τους λέει όχι, αλλά πρέπει να μάθετε να λέτε όχι. Γιατί, θα σας ρωτήσουν, γιατί γίνεται έρευνα κατά αυτού του ατόμου που είναι από το κόμμα μας. Εσείς θα πείτε ότι η έρευνα θα γίνει, δεν θα δεχθείτε πίεση ή να σταματήσουν οι έρευνες. Χρειαζόμαστε ισχυρούς ανθρώπους, ισχυρά πρόσωπα που ε, θα σταματήσουν την πολιτική παρέμβαση. Ισχυρά πρόσωπα τα οποία θα τα φοβούνται και οι άλλοι για να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στον εισαγγελέα να κάνει τη δουλειά του. Τώρα το πού θα βρείτε αυτά τα ισχυρά πρόσωπα που θα μπορέσουν ε, να, αρνηθούν την άσκηση πιέσεων, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να βρείτε ανθρώπους ακέραιους και ισχυρούς για αυτές τις υψηλές θέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μόνικα. Δύο ε, συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Τέσσερις. Κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών, διότι θα καθυστερήσουμε. Τέσσερις σύντομες ερωτήσεις και να ακούσουμε μετά τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με την ερώτηση που έθεσε η Χάιντι Χαουτάλα δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει ε, τριετής αναβολή της επικύρωσης ε, της συμφωνίας. Είναι κάτι που συμπεριλαμβάνεται στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, Ουκρανίας. εξυπηρετεί την καταπολέμηση, τον αγώνα μάλλον για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ε, δικαιωμάτων. Η Ουκρανία είναι θύμα λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Ε, είναι όμως κάτι που συνδέεται με, και με την καταπολέμηση της διαφθοράς, διότι συχνά βλέπουμε ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακριβώς ε, γίνονται για να συγκαλυφθεί η διαφθορά. Και θα ήθελα να πω ότι συμφορώ με τον κύριο Σαμπούνιν, η μαφία αντιστέκεται. Ναι, όχι μόνο στην Ουκρανία, παντού. Υπάρχουν άνθρωποι που πίεσαν ε, να γίνουν μεταρρυθμίσεις ε, στην Ουκρανία. Είδαμε η νεολαία πόσο ήθελε να αποκαλυφθούν ε, οι πράξεις της κλεπτοκρατίας του του καθεστώτος και μάλιστα είναι ανησυχητικό που βλέπουμε περιπτώσεις όπως ε, αυτού του νέου και νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, φέρνουν τεράστια ευθύνη και θα πρέπει να υποστηρίξουν την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Και υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν, να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, αλλά και τον εισαγγελέα και όσους άλλους είναι διατεθειμένοι ε, να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε υιοθετήσει ψήφισμα για την ανάκτηση ε, των ε, περιουσιακών στοιχείων και αυτό αποτέλεσε παράδειγμα για οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί και η Ουκρανία να το χρησιμοποιήσει. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο θα, έχουμε, θα δημιουργήσουμε μάλλον μια επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά και όλους τους φορολογικούς παραδείσους. Η διαφθορά στη δική σας χώρα συνδέεται στενά με ε, την διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ε, οι εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία στην Αυστρία, στην Λετωνία, στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αφορά λοιπόν όχι μόνο την Ουκρανία, αφορά και εμάς. Και γι' αυτό σας λέω, σας παρακαλώ, δώστε μας ό,τι στοιχεία έχετε, διότι το σύστημά μας, το χρηματοοικονομικό μας σύστημα χρησιμοποιείται ως σύστημα ξεπλήματος ε, χρήματος, ε, νομοποίησης παράνομων εξόδων. Και ο, ο, ο ε, κύριος ο πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Διαφάνεια, μόλις επισκέφθηκε την Ουκρανία και ελπίζω κύριε Λουτσέγκο να ε, δεχτείτε την προσφορά του, διότι και η Ουκρανία, όπως ε, και κάθε άλλη χώρα σε τέτοια θέση, χρειάζεται πολύ βοήθεια από όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ κύριο Σάιρος Βόλσκι. Δεν θα θέλω απλά να θυμίσω τη συζήτηση που είχαμε σήμερα, να σας ε, μιλήσω σήμερα για τη συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών για τη χορήγηση ε, δυνατότητας ε, μετάβασης στην Ουκρανία άνευ θεωρήσεων. Αυτό ήταν ένα σημείο καμπή το σχέδιο για τη κατάργηση των θεωρήσεων. Εγώ σύστησα όσο γίνεται πιο γρήγορα και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη χορήγηση αυτού του καθεστώτος. Αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ουκρανία να εξακολουθήσει να καταπολεμά την διαφθορά. Και για να την ενθαρρύνουμε ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια και για να βοηθήσουμε αυτές τις δυνάμεις που τη στηρίζουν τη διαφθορά, προτείνουμε το εξή. και παραθέτω τέσσερις σειρές της γνωμοδότησης για αυτό το θέμα. Φαντάζομαι θα γίνει δεκτή από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και από το Κοινοβούλιο στη συνέχεια. Για να μπορέσουμε περισσότερο να εθαρρύνουμε τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολουθήσεως που θα εξασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει δυνατότητα μόχλευση εφόσον συνεχίζεται η μεταρρύθμιση κατά της διαφθοράς και υπέρ της νομοθεσία υπέρ του κράτου δικαίου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν θα λειτουργήσει μόνο τώρα, αλλά θα συνεχίσει να ελέγχει. Τώρα όσον αφορά την χορήγηση, την κατάργηση του καθεστώτος βίζας, το ε, ε, ορεινός μηχανισμός αναστολής δεν αρκεί γιατί εστιάζεται μόνο στους κινδύνους μετανάστευσης ε, και θα πρέπει να συμπληρωθεί από την προσθήκη διαρκούς τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών και οροσίμων. Αυτό σημαίνει ότι προτείνουμε μια άλλη νομοθεσία που θα προσθέτει ότι η συνεχιζόμενη εφαρμογή και πρόοδος στους όρους που περιλαμβάνονται στη ΛΑΠ και στους όρους του IMF για την ε, Ουκρανία θα καταγραφούν ώστε να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε και να πιέζουμε ε, για να εκκριζώσει τελείως επιτέλους η Ουκρανία την ε, διαφθορά από τη δημόσιο βίο της. Ευχαριστώ. σμάκερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέη. Καταρχά, να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ που ήρθαν ε, σήμερα και μα έδωσαν πολύ ενδιαφέρουσε ε, πληροφορίε ε, και επίση και για τη ρουμανική υπόθεση και εμπειρία. Εγώ δεν είμαι μέλο αυτή τη επιτροπή, αλλά είμαι μέλο τη επιτροπή. Της Επιτροπής Συνεργασίας. Οπότε παρακολουθώ την τις εξελίξεις στην Ουκρανία εδώ και κάποια χρόνια. Είμαι Φλαμανδός, δηλαδή προέρχομαι από το δυτικό μέρος της Ένωσης. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ όμως για την Ουκρανία και στηρίζω τις μεταρρυθμίσεις. Η δικαστική μεταρρύθμιση είναι πολύ σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας στη χώρα μέσω της ανάπτυξης ενός δικαστικού συστήματος δικαίου, αποτελεσματικού, ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό στην καταπολέμηση εγκληματικότητα. Θα πρέπει να είναι αδιάφθορο και υπόλογο σε θεσμικό και ατομικό επίπεδο και πάνω απ' όλα θα πρέπει η κοινωνία να το εμπιστεύεται. Και ο κύριος Σαμπούν είναι και πάλι μίλησε για αυτά που και εγώ συναισθάνθηκα και έμαθα κυρίως την τελευταία μου επίσκεψη στην Ουκρανία πριν από μια-δύο εβδομάδες. Το είπα και στα σχόλιά μου μετά από τον πρώτο γύρο μιλωτών ότι είχα την αίσθηση ότι πολλοί κόσμοι έχει την εντύπωση πως το παλιό σύστημα αντεπιτίθεται, ότι το κατεστημένο μπόρεσε να, μάλλον ότι στη Μεϊντάν κατάφεραν να το κλειδονίσουν το κατεστημένο αλλά όχι να το ε, καταρρύψουν, όχι να τον κρεμίσουν. Αυτή την αίσθηση έχει ο κόσμος και ο χρόνος ε, δεν είναι σύμμαχος ε, σε αυτή την υπόθεση. Συμφωνώ μαζί σας ότι η πολιτική και ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ελίτ αντιπιτίθεται Και εγώ είμαι πολιτικός, αλλά για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη θα περίμενε κανείς οι πολιτικοί να πιέσουν για τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα ανέμενε κανεί για να μπορέσει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Για να αποφύγει ακόμα ένα νέο Μαϊντάν. Αντί να χρησιμοποιεί, να, να, να πατάει τον γκάζι και από την άλλη πλευρά να τραβάει το χειρόφρενο. Αυτό εμένα μου φαίνεται τρελό. Μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτή ε, ε, ε, η κατάσταση, πού οφείλεται, από πού έρχεται η πίεση. Ναι, πείτε μας ειλικρινά, από πού προέρχεται αυτή η πίεση, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, ποιανού συμφέροντα είναι τόσο μεγάλα ώστε να το κάνει αυτό. Και μια ευθεία ερώτηση προς τον κύριο Λουτσένκο. 5.000 χιλιάδες κερδίζει ένας ε, ε, υψηλό ιστάμενος δημόσιος Δηλαδή 180 ευρώ το μήνα. Πώς θα εμποδίσετε τη διαφθορά στο μέλλον όταν ο εισαγγελέα πρέπει να ζήσει με ένα τέτοιο μισθό τόσο χαμηλό. Πώς θα εξασφαλίσετε δεν θα συνεχιστεί έτσι η ίδια ε, κατάσταση, εφόσον ε, πηγή της διαφθοράς ε, πολλές φορές είναι η πολύ χαμηλή μισθή των δημοσίων υπαλλήλων. Τα λεφτά δεν είναι το παν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές τις πληροφορίες έχω εγώ, θέλω να ξέρω αν αληθεύουν όλα αυτά. Και πολύ ελπίζω ότι θα μεταρρυθμιστεί το δικαστικό σύστημα, γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη, στο κράτος δικαίου και πιστεύω και στην Ουκρανία. Τελευταία ερώτηση. Ελένα Πριστάνια από το ε, Ουκρανική δεξαμενή σκέψη ε, που βασίζεται εδώ, εδράζεται εδώ στην ε, Βρυξέλλα. Καταρχά, οι Ουκρανοί ε, υπάλληλοι και το, το, κοινό μιλάει για τις μεταρρυθμίσει, στους πιο δύσκολους τομεί του δικαστικού σώματος και το γραφείο του εισαγγελέα. Ε, και πραγματικά ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσουν και συνεργαζόμαστε μαζί σας. Ελπίζω ότι εδώ απεχώ και όσους έθεσαν τις ερωτήσεις ε, για την πίεση που ασκείται και την αντίσταση του συστήματος. Θέλω προσωπικά να ρωτήσω τον κύριο Πετρένκο και τον κύριο Λουτσένκο ποια είναι η προσωπική σας εμπειρία από την αντίσταση του συστήματος και πώς ε, εσείς αντιστέκεστε. Κύριε Πετρένκο, έχετε, είστε σε αυτό το αξίωμα εδώ και κάποιο καιρό και κύριε Λουτσέγκο πώς σκοπεύετε να ε, αντισταθείτε στο σύστημα. Ευχαριστώ. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον Υπουργό, δύο λεπτά, μετά ο κύριο Λουτσέγκο και μετά οι υπόλοιποι. Οι διερμηνήσεις έτσι και αλλιώς πρέπει να φύγουν σε δέκα λεπτά, γι' αυτό σας δίνω δύο λεπτά στον καθένα μόνο. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολιτική βούληση και για την ε, προσωπική σας στάση. Στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης βρίσκομαι δύο χρόνια. Ένα Υπουργείο παλαιομοδίτικο, παλαιού στυλ. Μεγάλη διαφορά στο σύστημα και σε πολλούς τομείς του Υπουργείου. Στο σύστημα καταγραφής ε, και μητρώου αυτοκινήτων ε, σε, πολλά, ε, σε όλους τους τομείς. Και ως υπουργό τι μπορεί να κάνει κανείς και στα πιο απλά πράγματα τι μπορεί να κάνει, να αλλάξει τα πάντα μόνο. Μέσα σε δύο χρόνια μειώσαμε δύο φορές το προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όταν ξεκίνησα είχαμε 27.000 υπαλλήλους. Τώρα έχουμε μόνο 12.000 υπαλλήλους. Όλα τα τμήματα όπου υπήρχε διαφθορά τα καταργήσαμε. Τις λειτουργίες τους τις αναθέσαμε είτε σε τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης είτε σε ιδιώτες. Ανοίξαμε όλα τα μητρώα, θεσπίσαμε νομοθεσία κατά της διαφθοράς που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Και όσον αφορά το πρόβλημα με το δικαστικό σύστημα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Οι δικαστές ήταν ανεξάρτητοι, αλλά είχαν τα ίδια προβλήματα με όλα τα άλλα συστήματα, όπως δηλαδή οι εισαγγελείς, οι αστυνομικοί. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το μεγαλύτερο μέρος του δικαστικού συστήματος και είναι μοναδική αυτή η ευκαιρία που μας δίνεται. Με τους ανοιχτού διαγωνισμούς, με τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των νομικών, της νομικής κοινότητας, μέσω των εγγυήσεων για την ανεξαρτησία των νέων ανθρώπων που θα μπουν στο σύστημα, μέσω των μισθών που θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, εξηγώντας σε αυτούς τους δικαστές ότι η ανεξαρτησία για αυτούς είναι υποχρέωση και ότι αν ε, διαπράξουν κάποιο αδίκημα και αυτοί θα πάνε στη φυλακή όπως οι άλλοι πολίτες. Δεν είναι δηλαδή μια ιερή κάστα πολιτών που βρίσκεται στο απειρόβλητο. Το παλιό σύστημα που δεν ήθελε να αλλάξει ανήκει πλέον στο παρελθόν. Τώρα δημιουργούμε ένα νέο σύστημα δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λουτσέγκο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Προς την κυρία Μακοβέη θέλω να πω ότι έγραψα στην παρουσίασή μου κρατική μαφία του Γιαννουκόβιτς. Το έχω γράψει. Και θέλω και να το εξηγήσω. Μου λένε συχνά, δεν μπορεί να συνεχίζεις να καταδιώκεις τον Γιαννουκόβιτς. Θέλω όμως να καταλάβετε ότι η ρίζα της αντιπολίτευσης σήμερα από αυτό ξεκίνησε. Αν έχω στα χέρια μου καταλόγους με σκάνδαλα του Γιαννουκόβιτς, και αν εξαγόραζε ψήφους βουλευτών με 2 και 3 εκατομμύρια, όπου και να κοιτάξετε, υπήρχε διαφθορά αν δεν καταδικάσουμε το σύστημα Γιαννουκόβιτς θα συνεχίσουν παντού και στο φορολογικό σύστημα και στα δασαρχεία, παντού θα συνεχίσουν να είναι διαφθαρμένοι. Θα νομίζουν όλοι ότι συνεχίζουμε ακριβώς όπως ήταν στο παρελθόν πασπαλίζοντας λίγο την επιφάνεια με έναν αέρα διαφάνειας. Συνεχίζει να υπάρχει το παλιό σύστημα. Και τώρα συνεχίζει και την περασμένη εβδομάδα ανακαλύψαμε κάποιους που είχαν καταχρεστεί ένα εκατομμύριο. Κάποιοι διέφυγαν στη Μόσχα, αλλά κάποιοι ακόμη βρίσκονται στην Ουκρανία και συνεχίζουν την πρακτική τους. Προσπαθούν να συνεχίσουν την επεξαίρεση χρημάτων. κατ' το σύστημα Γιαννουκόβιτς είναι διαπλεκόμενο με το σύστημα ε, ε, της διοίκησης και γι' αυτό μίλησα για την κρατική μαφία του Γιαννουκόβιτς. Πρέπει λοιπόν το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα να ασχοληθεί με τις παλαιές υποθέσεις. Οι καινούριε υποθέσεις θα είναι αντικείμενο του ΝΑΜΠΟΥ, του νέου γραφείου για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εμείς έχουμε την άμεση υποχρέωση να καταπολεμήσουμε τα παλαιά δικήματα. Και ως προς το ερώτημα του πώς θα τα καταφέρουμε, η απάντηση είναι ότι δεν θα φοβηθούμε. Εγώ έχω περάσει δύο Μαϊντάν, έχω περάσει φυλακή, έχω δει πόλεμο. Και ξέρω ότι μία είναι η συνταγή. Να μην υποκύψουμε στο φόβο. Να κάνουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε και θα πετύχουμε. Θα υποβάλω όλα τα στοιχεία που έχω για τις εγκληματικέ οργανώσεις και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την καινούργια κυβέρνηση, αλλά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, τρεις προκλήσεις υπάρχουν για τους Ουκρανούς ε, συναδέρφους μας. Καταρχάς, την εφαρμογή πολύ παλαιών αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση ή σχεδίων δράσης που ήδη έχουν εγκριθεί. η σχεδιων δρασης που ηδη εχουν εγκριθει στην ε, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Ε, δεύτερον, ε, έρευνες που να προσανατολίζονται στα αποτελέσματα. Θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες αυτές και τα στοιχεία να διαβαστούν στα δικαστήρια. Το κοινό περιμένει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, έχουμε πολλές παράνομες δραστηριότητες οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν. Και η άλλη πρόκληση είναι ο χρόνος, διότι ο λαός της Ουκρανίας έχει χάσει την υπομονή του τώρα πια. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει πολιτική λογική στον τρόπο που η ελίτ της Ουκρανίας ε, αντιστέκεται στις ε, μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν έχει καμία λογική κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον που βρισκόμαστε σε πόλεμο και οι άνθρωποι, οι πολίτες ε, δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν άλλοι. Ε, το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο πολιτικό. Η λογική που επικρατεί είναι οικονομική και διαφθαρμένη. Και κάτι ακόμα. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς έρευνες ή εργαλεία επιβολής του νόμου. Υπάρχουν διεφθαρμένα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, της ε, Κεντρικής Επιτροπής ε, Διορισμού των ε, Δικαστών. Αλλά όπως υπόθηκε, όλοι μπορούν να αλλάξουν, να αλλαχτούν με την πολιτική διαδικασία. Από τον πρόεδρο δηλαδή, από το κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία λογική που περιμένουμε και οι άνθρωποι αυτοί παραμείνουν στις θέσεις τους. Η πρώτη λοιπόν λογικά πολιτική κίνηση θα ήταν να τους διώξουμε από το σύστημα. Ούτε καν στη φυλακή δηλαδή, μόνο από το σύστημα να τους βγάλουμε. Και μετά σε δεύτερη φάση να πάνε στη φυλακή. Δεν καταλαβαίνω γιατί παραμένουν στη θέση τους όλοι αυτοί. Η κυρία Μακοβέλη, ευχαριστώ.